La séance est ouverte. Je voudrais vous indiquer mon intention d'ajouter deux points à l'ordre du jour. Ils viendront en discussion. Καλησπέρα σας. Στο τέλος της συνεδρίασης θα μιλήσουμε για τα διάφορα. Πρώτα απ' όλα, ε, Γενικός Εισηγητής για το 2016, τον προπολογισμό του 2016, ο κύριος Φερνάντες. Θα θέλαμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα 18 ε, εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, το σχετικό έμβασμα. Θα θέλαμε να μάθουμε λίγο περισσότερες πληροφορίες, κάτι το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε περισσότερα για την εφαρμογή αυτής της ε, διευκόλυνσης. Δεύτερο θέμα αφορά την ε, ανακοίνωση της, ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μας πει διευκρινήσεις ε, για ε, την ανακοίνωση της 7ης Ιουνίου σε σχέση με ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο της ε, ευρωπαϊκής ατζέντα ε, για τη μετανάστευση. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στο τέλος της ε, συνεδρίασης υπό τα διάφορα. Όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, υπάρχουν παρατηρήσεις. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται. Θα σας ενημερώσω τώρα για τις ε, αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές σήμερα το πρωί. Σε σχέση με την αποστολή που είχαμε προγραμματίσει στην Ελλάδα, καταρχάς για τις 18, ε, 19 και 20 Ιουλίου, αναβάλλεται σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία που θα την ε, επιβεβαιώσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, πρώτο εξάμεινο του 2017, αν επιβεβαιωθεί η αποστολή αυτή. Δεν θα την κάνουμε τον Ιούλιο γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί συμμετέχοντες. Δεύτερη απόφαση των συντονιστών θα ε, προταθεί να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης ε, διακοινοβουλευτικής μας ε, συνεδρίασης η θέση από κοινού των ε, εξωτερικών ε, συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνεργασία κατά περίπτωση με τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Ελέγχου του Προϋπολογισμού με σκοπό να είναι κάπως πιο ε, κοινά ε, τα δημόσια έξοδα, ε, όπως επίσης και οι συζητήσεις. Η κυρία Ολμέιερ για τη γνωμοδότηση την, για τη γνωμοδότηση που αφορά την, ε, τα δεδομένα εισόδου επικών τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την ε, υποβάθμιση των συνθήκων εφαρμογής του συστήματος εισόδου-εξόδου. Ε, ζητήσαμε από τον κύριο Ντεπρέ τη γνωμοδότηση για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον καθορισμό του κράτους μέλους που θα είναι αρμόδιο για την έγκριση της εφαρμογής ε, αίτησης ε, διεθνούς προστασίας από έναν από απάτριδες. Ε, επίσης, η ομάδα των σοσιαλδημοκρατών ε, για την ισότητα των φύλων και η κυρία ε, για τις οικονομικές δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2017. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα έχει μια έκτακτη συνεδρίαση στις 4 ε, Ιουλίου στο Στρασβούργο. Ε, και το για το 2017 και τον τριμερή διάλογο ε, για τις ε, πληρωμές θα αναβληθεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου λόγω του ότι ε, λάβαμε το σχέδιο προϋπολογισμού ε, με καθυστέρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα την ομάδα υψηλού επίπεδου για τους ιδίους πόρους, ε, θα λάβει χώρα στις 7 και 8 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας καλούμε να προσέλθετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, από κοινού με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών θα οργανωθεί ένα εργαστήριο για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και ε, της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά. Η, το εργαστήριο αυτό θα λάβει χώρα ε, στις 11 Ιουλίου από τις 4 στις 6.30 το απόγευμα και θα αφορά τις βελτιώσεις που μπορούν να υπάρξουν στον τομέα ε, της άμεσης ε, διαχείρισης. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας ε, πω ως ενημέρωση για τη συνεδρίαση των συντονιστών και τις σχετικές αποφάσεις. Επίσης τα πρακτικά της 11ης και της 25, 25 26ης Απριλίου σας έχουν υποβληθεί και αν δεν έχετε παρατηρήσει ως προς το περιεχόμενο των πρακτικών αυτών θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί επίσης. Πάμε τώρα το κύριο Όλμπριχ, το οποίος ε, έχει αναλάβει έκθεση που αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα διάφορα κράτη-μέλη. Κύριε Όλμπριχτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με την ε, ε απόφαση ε, του, με τη διάσκεψη, ναι, της, της των Προεδρών ε, ε, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με τη Ρέτζη γιατί προέρχεται από το 1B, τα χρήματα θα προέρχονται από το 1B που αφορά και την γεωργική πολιτική. λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την πολύ θετική ε, συνεισφορά τους, ειδικότερα για την Ελλάδα και την ε, Κύπρο για τις ε, οικονομικές προσαρμογές και βάσει αυτής της πολύ θετικής εμπειρίας η Επιτροπή πρότεινε να υπάρξει ένα πρόγραμμα για όλα τα κράτη-μέλη αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό θα γίνει σε εθελοντική βάση. Δηλαδή, αν, το, αν κάποιο κράτος μέλος το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει και αν γίνει αποδεκτό το πρόγραμμα βέβαια, τη στήριξη αυτή. Η στήριξη αυτή αφορά τεχνική στήριξη περισσότερο, συνεπώς ε, ε, επισκέψεις, ε, εκπαίδευση κλπ. Με σκοπό να ενισχυθεί ή να αναπτυχθεί η δυνατότητα ε, η διοικητική των διαφόρων ε, διοικήσεων, κυρίως όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν ε, είναι τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρξει ένας, μια άμεση σχέση ειδικότερα με το θέμα των ειδικών αναχώρα συστάσεων. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν λοιπόν παρουσιάσει τέτοιου είδους ε, ε, συστάσεις αναχώρα. Αν το κράτος μέλος ε, θέλει, μπορεί να ζητήσει αυτήν τη στήριξη για την τεχνική ε, βοήθεια. Προέρχεται από την πολιτική συνοχή που βρίσκεται τώρα στον προπολογισμό της Επιτροπής και μπορεί να ζητήσει τεχνική στήριξη και από το ε, πρόγραμμα ε, αγροτικής ανάπτυξης που βρίσκεται στον προπολογισμό της Γεωργίας. 142,8 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό και αυτό Από αυτά τα 112 προέρχονται από την τεχνική στήριξη και τα διαδοτικά ταμεία και 30, εκατομμύρια από την τεχνική στήριξη από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συνδέεται με τις ειδικέ αναχώρασης τάσης, ε, όπως είπα, και δεύτερον ότι είναι εθελοντική βάση. Το ερώτημά μου τώρα προς το, την Επιτροπή και προς τον Επίτροπο κατά τη διάρκεια της ακρόασης ήταν τι γίνεται στην περίπτωση που το, κράτης με, το κράτος μέλος ε, έχει λάβει τη σύσταση γι' αυτό, αλλά δεν θέλει να συμμετέχει σε τέτοιου είδους ε, στήριξη. Ποιες είναι οι συνέπειες, αλλά δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση, οπότε Συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω ότι έχουμε προετοιμάσει το πρόγραμμα αυτό. Το κείμενο μπορεί να τροποποιηθεί στις αρχές ε, του Σεπτέμβρη. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο ε, της διαδικασίας, αλλά βέβαια στην ε, περιγραφή του προγράμματος αναφέρονται διάφοροι τομείς πολιτικής. Είναι πάρα πολύ ευρύ το πρόγραμμα αυτό. Αφορά την επιχείρηση, την εκπαίδευση, τη μετανάστευση, διαφόρων ειδών πολιτικές και μια διαφορετικού είδους ε, ε, διαχείριση. Είναι διαφορετικές οι δράσεις που είναι επιλέξιμες, σεμινάρια, ε, εργαστήρια. Συνολικά 142 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Όλμπριχτ. Ποιο θα ήθελε να λάβει τον λόγο, ο κύριο Μάγκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και συμφωνώ μαζί του ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν μεγάλα προβλήματα για να εφαρμόσουν αυτήν την μεταρρύθμιση ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτή την ικανότητα σε διοικητικό επίπεδο για να μπορέσουν να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια βελτίωση και των οικονομικών μέσω αυτής της μεταρρύθμισης. Θυμόμαστε τον Ιούλιο του 2015 όταν ζητήσαμε από την Κομισιόν να έχουμε μία έκθεση για, τις, ε, για τα ποσά τα οποία δεν είχαν εκταμιευτεί, τα λεγόμενα RAL, για τα προηγούμενα τρία χρόνια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη σε σχέση με τα θέματα αυτά των διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων. Αν τελικά ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την διοικητική ικανότητα των χωρών αυτών, θα πρέπει τα κράτη-μέλη αυτά να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και το τοπικό επίπεδο, να μπορέσουν οι δήμοι, οι κοινότητες και οι πολίτες να συμμετάσχουν στην επίτευξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μαραγάλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον κύριο Όμπριχτ, πράγματι μπορούμε να εργαστούμε επί της βάσης που έχει παρουσιάσει. Εμείς έτσι κι αλλιώς μια γνωμοδότηση θα δώσουμε προς την Επιτροπή ΡΕΤΣΙ Περιφερειακών Θεμάτων. Πρέπει λοιπόν να εκφράσουμε την απόψή μας για αυτά τα 140 εκατομμύρια για την τεχνική αρρωγή. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για ένα θέμα που είναι καθαρά τεχνικό δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο λειτουργικού χαρακτήρα. Υπάρχουν ορισμένα θέματα ουσίας και γενικής ε, σύλληψης για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Μεταρρυθμίσεις προς ποια κατεύθυνση, για να πετύχουμε τι, για να ακολουθήσουμε ποιο υπόδειγμα. Ποια είναι η κοινή ευρωπαϊκή αναφορά η οποία εφαρμόζεται και σε ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται. Όλα αυτά μας φέρνουν σε μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει για να θεσπίσουμε κάποια κριτήρια για το πώς θα εφαρμόσουμε αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις. Ο Καν δεν ασχολήθηκε με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά είπε ότι για, για να ισχύει ένα υπόδειγμα θα πρέπει να είναι ε, να μπορεί να είναι επαληθεύσιμο, να μπορεί να ε, λειτουργήσει σε παραπάνω από μία περιπτώσεις. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να καταλάβουμε σε ποιο βαθμό εμείς μπορούμε να απαρνηθούμε τις αρχές της επικουρικότητας και να αφήσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να περιορίζεται σε μονάχα περιπτώσει κακοδιαχείρισης των πόρων, σε δευτερεύοντα αποτελέσματα μπορούν να αναπτύξουν άλλες χώρες για άσκηση πολιτικής dumping ή άλλων πολιτικών που δεν συνάδουν με την πολιτική ανταγωνισμού. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να έχει νόημα αυτό. <clears throat> Οι αρχές αυτές, προς το παρόν από ό,τι εγώ βλέπω, δεν περιλαμβάνονται στο μυαλό και στην αντιμετώπιση της Κομισιόν. Η Κομισιόν θέλει να προωθήσει ορισμένου στόχου όπω είναι η ιδιωτικοποίηση. Καλή ιδιωτικοποίηση. Αλλά έχουμε και αρνητικέ εμπειρίε από όλα τα κράτη-μέλη μα. Έχουμε κάποια ιδιωτικά μονοπόλια τα οποία μετά είχαν ακόμα χειρότερο αποτέλεσμα από ότι τα δημόσια μονοπόλια τα οποία καταδικάσουμε με τόσο μεγάλη ευκολία. Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων είναι ότι η εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα εφαρμόζονται με ένα μονοδιάστατο τρόπο προς μία μοναχα κατεύθυνση. Οι χώρες που έχουν έλλειμμα θα πρέπει να καλύπτονται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά όχι βέβαια οι χώρες οι οποίες έχουν πλεόνασμα, ακόμα και αν είναι σκανδαλωδόν δια, διαστάσεων αυτό το πλεόνασμα. Μιλάμε επίσης και για την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των κρατών μελών, αλλά αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι υποστηρίζουμε πολιτικές φορολογικού ντάμπινγκ και έχουμε εξόφθαλμες περιπτώσεις όπως αυτή της Ιλλανδίας ή το των κατοχωρών. Επομένω, έχει σημασία να έχουμε ένα κοινό μοντέλο επί του οποίου να βασίσουμε οποιαδήποτε αξιολόγηση που κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Μάργα. Μα δεν τελείωσα κύριε Πρόεδρε. Μία τελευταία φράση. Για να καταλάβετε πολύ καλά. Δεν λέμε όχι στην έννοια των διαχωτικών ε, αλλαγών και την ανάγκη μιας τεχνικής αρρωγής προς την κατεύθυνση αυτή. Πρέπει όμως να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και να βελτιώσουμε την κακή ή ανεπαρκή χρήση των διαδοτικών πόρων όπου χωρεί. Αλλά αυτή τη στιγμή η προσήγηση που έχουμε δεν είναι κατάλληλη να επιτύχουμε όλα αυτά. Αυτή η συζήτηση είναι συνδεδεμένη με άλλα θέματα όπως η μεταρρύθμιση του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου και η ικανότητα συλλογής εσόδων, θα πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε από κοινού. Λοιπόν, αγώνας κατά των ε, φορολογικών διακρίσεων και της βελτιστοποίησης σε φορολογικό επίπεδο. Υπάρχει αυτό, το οποίο το επιτρέπουν τα ευρωπαϊκά κράτη με την πολυμορφία των ε, κανόνων στο φορολογικό επίπεδο και τα λεγόμενα tax rulings. Αλλά δεν είναι μόνο πολυεθνικέ εταιρείε οι οποίε παίζουν αυτό το παιχνίδι για τον αγροτικό τομέα μπορώ να σα παρουσιάσω πολλά παραδείγματα φορολογική βελτιστοποίηση μέσα σε εισαγωγικά οι οποίε στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μέσα στην ίδια την ενία αγορά. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ενδιαφέρον θέμα όχι για την Επιτροπή Προπολογισμών αλλά ίσω και για κάποιου άλλου στο Κοινοβούλιο. Ντόνανο. Εγώ συμφωνώ με, σε μεγάλο βαθμό με αυτά που λέει ο κύριο Μαραγκάλ γιατί εδώ έχουμε μπροστά μας μια έκθεση που θα πρέπει να θέσει και το ερώτημα του τι μοντέλο θέλουμε να έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς θέλουμε. Μια ένωση η οποία είναι υπερφιλελεύθερη, όπως φαίνεται να ισχύει σήμερα, ή αντίθετα θέλουμε να έχουμε ένα μοντέλο το οποίο να είναι καλύτερα αριθμισμένο, το οποίο θα επιτρέψει στους πολίτες να είναι σε καλύτερη κατάσταση οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις είναι ένα ερώτημα ουσίας το οποίο τίθεται τώρα. Δεν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα σχήματος και τρόπου. Βεβαίω να υπάρχει μια βοήθεια στα κράτη τα οποία θέλουν να προβούν σε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, αλλά ακολουθώντα ποιο μοντέλο. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. <clears throat> και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε εμείς ποιο είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο. Επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο κ. Μαραγκάλ εμείς έχουμε τονίσει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική πτυχή και τη δημοσιονομική πτυχή. Αλλιώς δεν μπορούμε να φτάσουμε στην ουσία του προβλήματος. Ποιο μοντέλο και ποιο είναι το καλό μοντέλο, λέει ο πρόεδρος. Ναι, πράγματι. Μα είναι πολιτικό πρόβλημα αυτό, κύριε πρόεδρε. Μα είναι το σωστό μοντέλο είναι αυτό το οποίο οδηγεί σε ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, <clears throat> οδηγεί σε εξισορροπημένα οικονομικά, αυτό το οποίο οδηγεί στην πλήρη απασχόληση. Μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη βέβαια οικονομία. Αυτό είναι ένα καλό μοντέλο, αυτό είναι το μοντέλο το οποίο πρέπει να έχει η Ευρώπη, πιστεύω, λέει ο Του, του δεν θέλει κανείς να λάβει το λόγο. Ίσως μπορεί να κλείσει ο κύριος Όλμπριχτ. Δύο στοιχεία νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά και οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης που θα πρέπει να εμπλακούν και να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους προγράμματα. Όπως μας λέει όμως η Κομισιόν, ο μόνος τρόπος να εμπλακούν οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι μέσα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η ιδέα είναι το πρόγραμμα δίνει λεφτά στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη μετά έχουν τη δυνατότητα να το αποκεντρώσουν σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο δεύτερο στοιχείο. Πρέπει να πω ότι όλοι μας εκπλησόμαστε λιγάκι, γιατί το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο ήδη έχει καθοριστεί βάσει των συστάσεων αναχώρα. Υπάρχουν συστάσεις για το ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Και φυσικά αυτό προϋποθέτει ένα μοντέλο και αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο, είναι μια διαδικασία η οποία συνεχίζει εδώ και κάποιο διάστημα. <clears throat> Τώρα όμως είπαμε ότι αν τα κράτη-μέλη έχουν μια σύσταση για να κάνουν διαφορετικές αλλαγές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια για να εφαρμόσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να πούμε ότι δεν είναι μονάχα για χρήματα και τεχνική αρρωγή, αλλά ίσως θα πρέπει σήμερα να εγείρουμε το ερώτημα τι ακριβώς έχει προταθεί στα κράτη-μέλη και από πού προέρχονται τα χρήματα και σε τι είδου αλλαγέ προορίζονται. Τίποτα από αυτά δεν είναι σε αυτό το έγγραφο. Αυτό είναι πάρα πολύ τεχνικό. Λέει ότι μπορείτε να πάρετε λεφτά επί τη βάση των ειδικών αναχώρα συστάσεων με στόχο τι ε, διαφορετικέ αλλαγέ. Το έγγραφο λέει πώ θα πάρετε λεφτά, πόσα λεφτά μπορείτε να πάρετε, γιατί μπορείτε να τα πάρετε, πάντα σε εθελοντική βάση. Μα το ερώτημα πάντα τίθεται αυτό που είπε ο κ. Μαραγκάλ. Ένα ενιαίο μοντέλο, πολλά μοντέλα. Πώ μπαίνουν σε αυτά οι συστάσει και τι συστάσει παίρνουν τα κράτη-μέλη. Και ποιο προτείνει ποιο μοντέλο σε ποιο κράτο. Αλλά ίσως μπορούμε να δούμε να, ότι αυτό το έγγραφο μπορεί να είναι και ένα πρόσημα, μια ευκαιρία, ένα έναυσμα να ασχοληθούμε και επί της ουσίας. Αλλά καταρχήν αυτό το κείμενο είναι για το πώς θα πάρει κανείς τα χρήματα και πώς θα τα χρησιμοποιήσει η τεχνική αρρωγή. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε κύριε Όλμπρεχτ, να βγούμε από τον πέπλο τεχνοκρατικής υποψίας και να μπούμε σε ένα πολιτικότερο χώρο, αυτό θα είναι πολύ θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλα αυτά είναι συστάσεις της Κομισιόν. Θα ήταν καλό οι συστάσεις αυτές να μπορέσουν να <clears throat> έχουν και ένα πολιτικό υπόβαθρο. Δηλαδή ότι εμείς απλώς θα κάνουμε τον έλεγχο σε νομικό επίπεδο. Εγώ προσωπικά, λέει ο κ. Σόλμπριχτ, εγώ ξεκίνησα πάντα από την αρχή με τις ε, συστάσεις για την Πολωνία, τη χώρα μου. Πρώτη φορά τα, τις είδα αυτές τις συστάσεις. Είναι πολύ τεχνικές αυτές οι συστάσεις. Μα το ερώτημα είναι αν αυτές οι ειδικέ αναχώρα συστάσεις αφορούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ή αφορούν τη διοικητική ικανότητα. <clears throat> Γιατί εδώ αν θέλουμε μονάχα να ενισχύσουμε την διοικητική ικανότητα αυτό είναι διαφορετικό από τις διαρθρωτικές ε, αλλαγές. Εντάξει, δεν θέλουμε σφάλματα στην εφαρμογή και τα λοιπά, θέλουμε πραγματική διοικητική ικανότητα, αλλά αν θέλουμε να κάνουμε διαρθρωτική αλλαγή, αυτό είναι ένα άλλο παπά Ευαγγέλιο. Και αν είναι εθελοντική η βάση, όπως λέμε, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Είναι ένα είδος βοήθειας αλλά ίσως ε, στην επεξεργασία αυτής της έκθεσης ίσως θα βρούμε κάποιες απαντήσεις για τα θέματα αυτά. Θα τα ξαναπούμε στην 1η Σεπτεμβρίου και οι τροπολογίε για την έκθεσή σας πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα στις 8 Σεπτεμβρίου, θα ψηφίσουμε στις 11 Οκτωβρίου και η έκθεση στην Επιτροπή Ρέτζη θα ψηφιστεί τον Νοέμβριο του 2016 και στην Ολομέλεια λίγο αργότερα, δεν ξέρουμε ακριβώ πότε. Η κυρία Γουάρδια Σαάλ για το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, έτσι, σωστά. Αφρική, Καραϊβική ειρηνικός σημαντική, μεγάλη περιφέρεια και η Ασία εκεί κοντά. Αυτό πρόκειται για ένα κείμενο για την Επιτροπή Ανάπτυξη όσον αφορά για το μέλλον των ισχυωσιών μας και για το τμήμα του προπολισμού που αναλογία. αναλογεί. Άπαξ και κλείσει το 2020 θα λήξει η Κοτονού Κατά σύμπτωση επίση έχουμε και τη λήξη του δημοσιονομικού πλαισίου, αυτό το οποίο ισχύει τρεχόντω. Οπότε και θα πρόκειται για μια υπέροχη ευκαιρία που θα έχουμε ούτω ώστε επιτέλου να μπορέσουμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη που τώρα είναι εκτός ε, να μπορέσουμε επιτέλου αυτό να το καλύψουμε στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι επομένω ε, ιστορική στιγμή αυτή για το Κοινοβούλιο και αυτό θέλουμε να καλυφθεί από αυτό από το δημοσιονομικό πλαίσιο και να αποκτήσει περισσότερη νομοποίηση και αποτελεσματικότητα η ενίσχυση και ταυτόχρονα να υπάρχει μια συνεχτικότητα, μια συνέπεια μεταξύ των πολιτικών που αναλογούν στα διάφορα ταμεία ε, και από την άλλη μεριά συνέπεια με τις άλλες πολιτικές της ε, Ένωσης. Έχουμε και κάποια άλλα ταμεία, κάποιους άλλους πόρους εκτός προϋπολογισμού. Ε, αυτά τώρα είναι κάποιο τρόπο της μόδας έρχομαι επομένω σε αυτό το περίφημο ημισονομικό πλαίσιο όπου και θέλουμε να εντάξουμε αυτή την υπόθεση, αυτή τη χρηματοδότηση. Ε, Επίση, θα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει εάν σκέφτεται να καλύψει από την μέλουσα προσεγή ε, απόφαση το Ταμείο Ανάπτυξη και έτσι να μας δώσει κάποιο χάρτη για το πώς θα πορευτούμε. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία. Είπαμε και για το καταπίστευμα για την Αφρική και έχουμε το κείμενο το οποίο εδώ πέρα εγκρίναμε και είπαμε ότι δεν θέλουμε να περικόψουμε χρήματα από άλλες πολιτικές. Δεν θέλουμε να κόψουμε από τα καταπιστέματα που έχουμε από ε, τα άλλα μέτωπα και φυσικά θα, πρέπει κάτι να κάνουμε όσον αφορά την εκπτώση της ε, φτώχειας και έτσι με έναν αποτελεσματικό τρόπο να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα των ε, εκτοποιήσεων προσφυγικό. Τέλος κάτι άλλο το οποίο το συζητούμε συνέχεια εδώ πέρα στην Επιτροπή είναι το πώς τα χρηματοδοτικά καινοτόμα μέσα θα μπορέσουμε να τα χειριστούμε και ίσως και να τα συνδυάσουμε με κάποιες ενισχύσεις, επιδοτήσεις όπου και σε κάθε περίπτωση να έχουμε την επιλογή ελεύθερη και έτσι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και την απόδοση να πιάσουν τόπο τα λεφτά μας δηλαδή για τις επιδόσεις μας για, να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος και δεν να θέλουμε επομένω να κόψουμε κάποιες ε, επιδοτήσεις, ενισχύσεις και να τις αντικαταστήσουμε με αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Και επομένως θα πρέπει να έχουμε ε, επιλογή εργαλείων για κάθε περίπτωση και κάτι άλλο. Έχουμε τώρα την ε, πρωτοβουλία της Κομισιόν, αυτή την πρόσφατη, αυτή την καινούργια ιδέα για επένδυση για την Αφρική, κάτι, κάτι σαν πλάνο Γιούγκερ για την Αφρική. Και επίση ε, σχετικά με αυτό να μα πει η Κομισιόν τι λέει. Μπορούμε εμεί ως Κοινοβούλιο δυναμικά και ενεργά να συμμετάσχουμε. Ε, ευχαριστώ λέω πρόεδρο. Πλάνο Γιούγκερ για την Αφρική. Η κυρία Μογγελίνη έκανε κάποιες ανακοινώσει πριν εβδομάδα σχετικώ. Ε, τότε τότε θα πρέπει να δούμε πώς ο προϋπολογισμός θα δώσει λύση για το μεταναστευτικό. Οπότε και ταυτόχρονα θα κάνουμε κάτι και για τις πηγές του προβλήματος. Άρα να βοηθήσουμε τους Αφρικανούς να αναπτυχθούν οι Αφρικανικές χώρες. Οπότε και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι όπως είπατε προπολογισμό να συνεχίσει να συνδυαστεί με το Ταμείο Ανάπτυξη. Και να έχουμε και αυτή τη με αξιολόγηση. Επίτευξη, επίτευξη σας τα λέω αυτά, είναι μια πρόκληση. Bon. Euh, Ποιος θα ήθελε τον λόγο σε σχέση με αυτά που μας είπε η κυρία Γκραντιοθάβολα. Ουδή. ε, ενός, ναι, νομίζω σημαίνει ότι ομονοούμε στις 15 θα γίνει η ανταλλαγή απόψε στο 22 μεσημέρι θα έχουμε την λήξη προθεσμία για κατάσταση τροπολογιών στις 11 Ιουλίου πρόκειται να ψηφίσουμε την έκθεσή σας κυρία Καρδιά Τσάπαλ στις 31 Αυγούστου η Επιτροπή Ανάπτυξη θα ψηφίσει το τελικό κείμενο και δεν ξέρουμε πότε θα κατέβει το κείμενο στην Ελλάδα Κύριε Αλή, είστε έτοιμος για να μας μιλήσετε για τα εργαλεία. Τα εργαλεία κατά της ασταθής των τιμών στις γεωργικές αγορές. Και βέβαια δεν είναι μόνο η αστάθεις των τιμών, αλλά θα πρέπει και οι τιμές να καλύπτουν τους αγρότες. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. είναι κοινά χαρακτηριστικά σε όλε τι αγορέ. Όμω πολλέ φορέ έχουμε μεγάλε διακύμανσει. Τα πράγματα οδηγούν στη στροφή τη μεγάλη αστάθεια. Οπότε υπάρχει πρόβλημα για του καταναλωτέ και του καταναλωτέ. Και πρόσφατα η παγκόσμια αγορά είναι μάρτυρα πολύ μεγάλων ασταθειών στι τιμέ των εμπορευμάτων και εκτινάχθηκαν οι τιμέ των τροφίμων και στα, σε, σε ύψη ρεκόρ από το 2008 οι τιμές των, ε, τροφίμων πέσαν το χειμώνα και ξανά μετά σήμερα ε, θεωρούμε ότι θα ισχύσει αυτή η αστάθεια των τιμών και για όλες τις γεωργικές αγορές και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια απειλεί για την διατροφική ασφάλεια. Ταυτοχρόνω, δε αυτού του είδου το ευμετάβλητο έχει να κάνει και με άλλες μεταβλητές μακροοικονομικές και αυτό οδηγεί σε ένα κακό περιβάλλον για τα υγειοργικά προϊόντα γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε προβλήματα και άρα με άλλους κλάδους όπως ε, την ενεργειακή αγορά. Βέβαια και αυτή η αστάθεια οφείλεται και σε διάφορα γεγονότα της παγκόσμια κοινή, οφείλεται στην, ε, στην αλλαγή του κλίματος και, και κάποια διαρκτικά άλλα προβλήματα για τις τιμές της ενέργειας, τις τιμές των λιπασμάτων, αλλά και τις συνταγματικές ισοτιμίες. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι η πρόταση μας ε, αφορά την Επιτροπή Γεωργίας επίσης και είναι εκείνη η αρμοδία επιτροπή ούτως ώστε να αγκαλιάσει αυτές μας τις προτάσεις για το ψήφισμα. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο παγκόσμιο εισαγωγέ και εξαγωγέ αυτών των γεωργικών προϊόντων και χρησιμοποιούμε τα προγράμματα για την ε, ΚΑΠ και για την ε, ε, Ήπεθρο ούτω ώστε να ενισχύεται το εισόδημα αλλά δεν έχουμε πετύχει ως αυτό το εισόδημα των αλλοτών. Θέλουμε να υπάρχει καλύτερη συνέργεια μεταξύ κάποια κάποιων των λοιπών πολιτικών ιδίω όσον αφορά την ε, ε, ενέργεια, τη χρήση της γης, την βιοπικιλία, τα οικοσυστήματα και επίσης να αναπτυχθούν οι μειονεκτούσες ορεινές και λοιπά περιοχές. Επίσης θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα για την προστασία του εισοδήματο των γεωργών και έτσι να μπορούν να αμείβονται οι προσπάθειες οι οποίες καταβάλλουν και έτσι να συμπληρωθεί η μεταρρύθμιση του 2014 με 20. Πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου παρακολούθηση τη αστάθεια των τιμών για τα γεωργικά προϊόντα και έτσι να βελτιωθεί το εργαλείο παρακολούθηση των ευρωπαϊκών ε, τιμών γεωργικών προϊόντων. Κύριε Αλή, ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Τι θέλει το λόγο σε σχέση με αυτό που ο κύριο Αλή. Monsieur Fernandez. Me pardonnera, Monsieur Donano. Oui, Monsieur le Président. Monsieur εύστοχη. Υπάρχει πρόβλημα σήμερα στην γεωργία λόγω της αστάθειας των ε, τιμών. Είναι δυνατόν να μένουμε στα βρωμένα χέρια προς αυτό το φαινόμενο. Χρειάζεται σταθερότητα υπέρ των γεωργών. Πολύ σημαντικό αυτό. Τη σημερινή ημέρα είναι μεγάλο ρίσκο να είναι κανείς γεωργός. Λόγω της αγοράς, λόγω του περιβάλλοντος, της πολιτικής έχουμε όλες αυτές τις ε, μεταβλητές. Ουδέποτε μπορεί να είναι σε ασφαλές περιβάλλον διάλογος. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάτσει και να εξασφαλίσει το εισόδημα των γεωργών. Άρα καλά τα λέει η έκθεση. Φυσικά και πρέπει και η κερδοσκοπία να χτυπηθεί όσον αφορά ε, τη Είναι πολύ κακή κερδοσκοπία, ακόμα χειρότερα όταν αφορά τα τρόφιμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Αλή για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι περίπου ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην θεσπίσουμε κάποιες καταστάσεις ως αμετάβλητες, κάτι το οποίο θα ισχύει για όλη την αιωνιότητα Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο προπολογισμό μας στο μεγαλύτερο μερίδιό του αφορά την γεωργία. Θα πρέπει να δούμε αν και στο μέλλον θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται κάτι τέτοιο. Και συζητήσαμε στο προηγούμενο σημείο της τη διάταξη ότι έχουμε και άλλες χώρες του κόσμου όπως είναι οι αφρικανικές χώρες που πρέπει να τις ενισχύσουμε και για να τις ενισχύσουμε θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν μια ανταγωνιστικότητα, το οποίο σημαίνει οι χώρες αυτές να μπορούν να εξάγουν προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αφορά σε μεγάλο βαθμό αγροτικά προϊόντα. Αν εμείς λοιπόν κάνουμε αυτούς τους κανόνες, θα πρέπει οι κανόνες μας να μην οδηγήσουν σε μια οχύρωση της αγοράς μας και μια αποτροπή των άλλων να εξάγουν προς την Ευρώπη, να βοηθήσουμε προφανώς τους γεωργούς, αλλά αυτή η αρρωγή προς τους γεωργούς δεν μπορεί να είναι χωρίς όρια. Θα πρέπει να θεσπίσουμε συνθήκες ανταγωνισμού, αλλιώς εμείς απλώς παγιώνουμε μία κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί και ξέρουμε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο σε 10 χρόνια κανείς δεν θα έχει τη θέληση να αλλάξει την πολιτική. Εδώ όμω θα πρέπει να δώσουμε και ένα μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά και, μια, και στην ευελιξία. Ο κύριο Μπέργκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε ο εισηγητής. Βρισκόμαστε σε μια δραματική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Όπως δεν έχουμε γνωρίσει για πολύ καιρό. Υπάρχει μεγάλη, διακύμα... μεγάλη διακύμανση των τιμών υπήρξε αυτή η περίοδος των βροχών που είχε κάποιες επιπτώσεις στην τιμή των προϊόντων και επομένως το εισόδημα των γεωργών. Αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε δει για δεκαετίες. Τώρα όμως έχουμε μια τόσο μεγάλη διάσταση στην ε, μεταβλητότητα των τιμών ώστε θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια άλλη δομή πέραν αυτής που είχαμε στο παρελθόν. Επομένως, τίθεται το ερώτημα πώς θα αντιμετωπίσουμε τον τομέα αυτό της γεωργίας και τις γεωργικές, τις περιοχές της υπαίθρου, τις αγροτικές που εξαρτώνται από τη γεωργία. Συμφωνώ με τον κύριο Ντονάνο λοιπόν ότι αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Ευτυχώς θα έλεγα έχουμε ένα σύστημα υποστήριξης του εισοδήματος των γεωργών μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Φανταστείτε αν αυτά τα εισοδήματα, τα οποία φυσικά υπόκειται σε κάποιες ε, προϋποθέσεις, αν δεν υπήρχε αυτή η εισοδηματική στήριξη. Το ίμιση και παραπάνω ίσως του εισοδήματος πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Γεωργία βασίζεται στις ευρωπαϊκές αρρωγές. Θα χρεοκοπούσανε όλοι λοιπόν. Επομένως προσοχή όταν μιλάμε για αλλαγές, όταν δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα πώς θα κινηθούν οι συνθήκες στη Γεωργία δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά βλέπουμε ότι τα, οι αρρώσιμες γέες και το νερό είναι όλο και πιο σπάνια και σε μεγαλύτερη ζήτηση και η δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων ορισμένων χωρών ίσως θα μπορούσαν να εξελιχθούν θετικά. Αν καταλάβουμε ποιες είναι οι πραγματικές τάσεις θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Όταν τώρα περάσουμε στο θέμα της πολιτικής ανάπτυξης, εδώ θέλω να σας υπενθυμίσω <clears throat> ότι δεν υπάρχει ένα εμπόδιο από την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε ήδη θεσπίσει τη στρατηγική Everything But Arms για τις πιο φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες, όλα εκτός από τα όπλα, για να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες. Έχουμε λοιπόν τις απαραίτητες ε, ε, δομές και θα πρέπει να δούμε αν είναι το σωστό αυτό που κάνουμε σε ε, επίπεδο αναπτυξιακής πολιτικής. Ακόμα και οι βοήθειε στον προπολογισμό των χωρών αυτών. Υπάρχουν πολλοί εδώ οι οποίοι δεν συμφωνούν με κάτι τέτοιο. Υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν προοπτικέ με τον τρόπο αυτό. Αλλά είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι καταδεικνύουν με μελέτε ότι για κάθε ευρώ που μπαίνει σε μια χώρα βγαίνουν 10 και πηγαίνουν στα Καϊμάνι στον Παναμά. Εδώ λοιπόν και η Κομισιόν θα πρέπει να πράξει τα απαραίτητα, γιατί είναι δική της αρμοδιότητα να υποβάλει προτάσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια αυξανόμενη, <clears throat> ένα αυξανόμενο ανταγωνισμό στην γεωργία και είναι και άνισες οι συνθήκες αυτού του ανταγωνισμού. Συγχρόνως υπάρχει τεράστια υπερσυγκέντρωση σε ό,τι αφορά τις αγορές τροφίμων. Πολλοί είναι, αυτή, είναι σε πολλές χώρες λίγες εταιρείες 4-5 που συγκεντρώνουν το σύνολο της ε, παραγωγής και της ε, διανομής και μάλλον της διανομής και της πώλησης και μόνο στην παραγωγή υπάρχει κάποια αυτονομία. Οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτή την υπερσυγκέντρωση των ε, επιχειρήσεων και των μονοπωλίων στον τομέα των τροφίμων. Είναι αυτό ουσιαστικά ανταγωνισμός ή ο μικρός γεωργός βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλες εμπορικές οντότητες τις οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και όταν πρέπει να κάνει ε, διαπραγματεύσεις για τιμές και να πρέπει να διαπραγματευτεί για έξι μήνες προηγουμένως πριν γίνει συγκομιδή, μετά από λίγο του λέει ο, ο έμπορος έχουν αλλάξει συνθήκες, αυτό που θα σου έδινα ένα ευρώ τώρα θα σου δώσω 80 cents. Αυτή είναι μια εμπειρία που γνωρίζουν πάρα πολύ στον γεωργικό τομέα. Αυτό δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση λοιπόν. Προφανώς είναι μια τεράστια προβληματική πρέπει να δούμε και δεν ε, θέλω να παραγνωρίσω και τη σημασία του να έχουμε νοπά και φρέσκα προϊόντα τα οποία δίνουμε στους ε, καταναλωτές. Αλλά το αν θα έχω γάλα σε μπλε ή σε πράσινο χαρτόνι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν τα μέτρα τα οποία έχουμε εμείς ε, εδραιώσει και θεσπίσει επιτυγχάνουν τους στόχους που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι επαρκή ή ανεπαρκή. Εάν όχι, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο είναι υγιής ή όχι η τωρινή κατάσταση στον τομέα της γεωργίας. και <clears throat> βλέπουμε ότι όταν γίνεται αυτή η διαδικασία του ντάμπινγκ από ορισμένου, αυτό θίγει όλη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και κυρίως το γερδό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οι προλαλήσαντες με κάλυψαν Είναι πολύ επικοδομητική η ατμόσφαιρα. Ε, ελπίζω να μεταφραστεί σε κάτι. Όσοι γνωρίζετε τη βίβλο θα ξέρετε ότι υπήρχε καλή επταετία και μετά κακή επταετία. Ας ελπίσουμε ότι θα... Δεν μπορούμε να ελπίσουμε μάλλον ότι επτά ε, συνεχή έτη θα είναι καλά στη Γεωργία. Στη δική μου χώρα είχαμε 26 χρόνια αρκετά ε, καλά και αν ένας γεωργός πτωχεύει συμβαίνει αυτό γιατί είτε πήρε κάποιο είδους κακές πιστώσεις είτε γιατί δεν ήταν αρκετά καλές οικονομικές του γνώσεις αλλά όχι επειδή δεν έλαβε υποστήριξη. Νομίζω λοιπόν ότι η υποστήριξη της Ένωσης προς τους ε, αγρότες ε, είναι πολύ αποτελεσματική. Αλλά το θέμα που πρέπει να θέσουμε σήμερα είναι το εξής. Ποια είναι η στρατηγική μας για έναν ορίζοντα 15 ετίας. Εμένα καθόλου δεν με ενδιαφέρει πώς θα αλλάξει η γεωργία μέχρι το 2020, γιατί θα είναι μόνο εν μέρη οι αλλαγές αυτές. Αυτό που με νοιάζει είναι πώς θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 2000, το 2030. Γιατί τα σημερινά μέσα που αποφασίζουμε θα έχουν αποτέλεσμα τότε. Ε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για τους αγρότες. Εγώ δέκα χρόνια είχα μία επιχείρηση και για τρία χρόνια ήμουν έτοιμος για πτώχευση γιατί δεν είχα ιδέα τι ακριβώς ε, γινόταν. Υπάρχουν ε, οι υποδηματοποιοί, οι οποίοι πάρα πολλές φορές πτώχευσαν μέχρι να χτίσουν τις τεράστιες ε, επιχειρήσεις τους. Ε, πράγματι, ξέρουμε, υπάρχει ξηρασία, υπάρχουν βροχοπτώσεις έντονες, συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, Προφανώς θέλουμε να βοηθήσουμε τη γεωργία, που είναι μία πτυχή, αλλά υπάρχει και το θέμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που είναι η άλλη πτυχή. Μετά το 2030 οι αγρότες πρέπει να είναι σε θέση να επιφέρουν κάποια προστιθέμενη αξία, για παράδειγμα στέγαση στο αγροκτημά τους. Αυτό σε μερικές ε, εκμεταλλεύσεις δουλεύει πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι λοιπόν η συνεισφορά μου στη συζήτησή μας σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να επενδύουμε τόσα πολλά κονδύλια της Ένωσης ε, για τη γεωργία μετά το 2030. Νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε καινοτομίες που θα επηρεάσουν και θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πλέον αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, ε, Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγχαρητήρια. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αλή για το σχέδιό του. Πιστεύω το κείμενο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε δύο ερωτήματα. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος μας προηγουμένως, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα μετά από την επιβολή του εμπάρκου στη Ρωσία, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δραματική κατάσταση στον αγροτικό τομέα και ιδίως στις αγροτικές αγορές. Αυτό αφορά ιδίως την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και το χείριο κρέας. Και αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη, είτε είναι παλιά μέσα σε αγωγικά, είτε είναι καινούρια. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές ότι αυτή η γνωμοδότηση δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα αυτά, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία προτείνονται για να αντιμετωπίσουν αυτή η κατάσταση έχουν κάποια προοπτική, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει και μία συμφωνία γενικά μεταξύ μας για να βγουν τα ποσά από την κοινή αγροτική πολιτική ώστε να στηριχθούν οι αγροτικές αγορές οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία. Επειδή ο πρόεδρος μας είναι και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, ελπίζω ότι θα δείξει κατανόηση για το πρόβλημα αυτό. Και ένα δεύτερο τώρα θέμα. <clears throat> Υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους γεωργούς για την υποστήριξή τους, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς. Αλλά στην πράξη αυτό μονάχα ισχύει και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με μονομένη γεωργία. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε και αυτό το σημείο. Γιατί αυτό δημιουργεί δυσκολίες στους γεωργούς, ιδίως σε μια δύσκολη εποχή όταν υπάρχουν όλο και περισσότερα καθήκοντα και υποχρέωσεις που επιβάλλονται στους γεωργούς, παραδείγματος χάρη ευμαρία των ζώων, το περιβάλλον, όταν έχουν υποχρεώσεις, όταν έχουν υποχρεώσεις οι οποίες αυξάνουν το κόστος παραγωγής, όπως είπαμε, για να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, πρέπει να καταλάβουμε το βάρος που υπάρχει και στο Γεωργό. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του καταναλωτή υπάρχει μια τεράστια πίεση ε, στις τιμές γιατί υπάρχουν οι εναλλακτικές πηγές από τις εισαγωγές προϊόντων τρίτων χωρών. Από τη μια μεριά λοιπόν αφήνουμε να μπαίνουν προϊόντα από τρίτες χώρες χωρίς, κανένα, χωρίς καμιά επιβάλληση, ενώ η γεωργοί μας και η παραγωγή των ε, ηθαγενών γεωργών επιβαρύνεται όλο και περισσότερο με υποχρεώσεις. Μαραγκάλ. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είμαι εμπειρογνώμων στα θέματα της γεωργίας, αλλά θέλω να καταθέσω μόνο μία σκέψη, αντιδρώντας σε όλα αυτά τα σχόλια που ελέγχθησαν, ιδίως του κυρίου Ντανόνα και του Ντανά, και τον κύριο Μπέγκερ, υπάρχει μια στρέβλωση λόγω της έννοιας <clears throat> της ε, ελεύθερης αγοράς που έχει εδραιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνουμε πολλές φορές σε κατάσταση μονοψωνίου από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ουσιαστικά ένα ολιγοπόλιο, ε, ένα ολιγοψώνιο ουσιαστικά στην αγορά αγροτικών προϊόντων. Αυτό το μονοπόλιο είναι λοιπόν σε θέση να ε, συμπεριλάβει στην πολιτική τιμό του την ε, παρουσία των αγροτικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο επιτρέπει στα ολιγοψώνια να επηρεάζουν την αγορά και ουσιαστικά να εμποδίσουν τους άλλους να μπουν στην αγορά. Αυτό κάνει πιο έντονη την υποχρέωσή μας πέραν του γεγονότος ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε έκτακτες συνδίκες της αγοράς που οφείλονται και σε αυτή τη στρέβλωση, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στρέβλωση της αγοράς. Ευχαριστώ. Εν ολίγης, θεωρούμε ότι βοηθούμε τους ε, παραγωγούς και ουσιαστικά οι καταναλωτές είναι αυτοί που παίρνουν τη βοήθεια αυτή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρεγκάλο. Κύριε Χριστοφόρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ορθά ο ευρωπαϊκός προπολογισμό χρηματοδοτεί και στηρίζει τον αγροτικό Δεν είναι τυχόν πω όλε οι χώρε του κόσμου και ιδιαίτερα ανεπτυγμένε όπω είναι οι ΗΠΑ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον αγροτικό τομέα. Όμως πρέπει να διαπιστώσω ότι σε αυτήν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχαν χώρες οι οποίες είχαν αυξημένο αγροτικό τομέα και σε δεικνώθηκαν και άλλες χώρες που μεγεθύστηκε ο αγροτικός του τομέας. Πιστεύω ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πάνε στοχευμένα. Και όταν λέω στοχευμένα, συγκεκριμένα υπάρχουν χώρες που έχουν συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα για συγκεκριμένα προϊόντα λόγω των καιρικών συνθήκων. Υπάρχουν άλλες χώρες που δεν τα έχουν πρέπει στοχευμένα να στηρίζουμε του τομεί εκείνου που μια χώρα στον αγροτικό τομέα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα με ανταγωνιστικά προϊόντα και όχι να δίνουμε αυτέ τι βοήθειε ουσιαστικά χωρί έλεγχο και χωρί στόχευση. Η χώρα η δικιά μου είναι μια από αυτέ που συρρυκνώθηκε ο αγροτικό τομέα. Όμω πιστεύω ότι έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και έπρεπε να στηριχθεί σε συγκεκριμένου τομεί που θα μπορούσε να κερδίζει και η χώρα μου και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με άλλε χώρε. Άρα πιστεύω ότι δεν φτάνει μόνο να λέμε ότι δίνουμε το 45% του προπολογισμού στον αγροτικό τομέα. Αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτε. Εάν αυτά τα χρήματα πραγματικά δεν έχουν και την ανάλογη απόδοση μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Σίγουρα το εμπάρκο της Ρωσίας δημιούργησε πολλά προβλήματα. Ε, πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς το διαχειριζόμαστε και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο. Γιατί στο τέλος με το εμπάρκο είναι ταπεινή μου άποψη ότι θα βοηθηθεί αγροτικά η Ρωσία. Γιατί την υποχρεώσαμε να επικεντρωθεί στον αγροτικό της τομέα, τον αναπτύσσει, ουσιαστικά προσπαθεί να γίνει αυτοδύναμη αγροτικά και στο τέλος είτε έχει εμπάρκο η Ρωσία είτε δεν έχει εμπάρκο, δεν θα χρειάζεται να εισάγει προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται διαχείριση λελογισμένη. Μπορούμε να βρούμε άλλους πολιτικούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία, αλλά ιδιαίτερα ο τρόπο που πλήττει το αγροτικό τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τη Ρωσία είναι πολύ σημαντικό θέμα και πιστεύω ότι πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ. Πράγματι, είναι, υπάρχει ιδιαιτερότητα στη γεωργία και υπάρχει βέβαια και ιδιαιτερότητα της κοινή γεωργικής πολιτικής που προφανώς δεν ε, εκπληρώνει την αποστολή της. Μέσα σε δέκα χρόνια οι Αμερικάνοι γεωργοί είδαν ε, το, τα έσοδά τους να αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό ενώ οι Ευρωπαίοι αγρότες έχασαν ε, σε σχέση με την αρχή της ε, περίοδου και αυτή η κοινή γεωργική πολιτική είναι ένας τρόπος για τα κράτη-μέλη να ε, λάβουν κάποια έσοδα ε, ως ανταμοιβή για τη συνεισφορά τους. Ε, τελικά βοηθάμε τη γεωργία σε μια χρονική στιγμή ε, που δεν έχει ανάγκη ή τη στιγμή ε, που οι τιμές είναι αρκετά υψηλές και υπάρχουν ε, βέβαια και υπάρχει και ο πειρασμός μεγάλα καταστήματα που έχουν ολιγοπόλιο και που έχουν κατάχρηση, που έχουν δεσπόζουσα θέση να, να ζημιώνουν τους γεωργούς υπέρ των καταναλωτών. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, ξανά να εξετάσουμε ξαναεξετάσουμε αυτήν την γεωργική πολιτική. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αλή. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ένα σύστημα εγγυήσεων κατά κάποιο τρόπο, όπως και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, αν όμως μειώθηκαν οι τιμές, αυτό συμβαίνει γιατί έχει αυξηθεί η παραγωγή. Πάρτε παράδειγμα το γάλα σε πολλές χώρες, όπως οι κατοχώρες και η Ιρλανδία για παράδειγμα, ξεκινήσαμε με αφετηρία το γεγονός ότι θα έπρεπε να ε, παράγουμε πολύ περισσότερο. Ε, τόσο μεγάλη παραγωγή σημαίνει μείωση τιμών σημαντική. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε και τον όγκο της παραγωγής, να μειώσουμε την παραγωγή για να μπορέσουν να αυξηθούν οι τιμές. Γιατί τώρα βρισκόμαστε σε μια μη βιώσιμη κατάσταση και οι παραγωγοί δεν μπορούν συνέχεια να πουλούν και να χάνουν, να έχουν ε, ζημία. Αυτό είναι ένας ε, ε, φυσικός νόμος. Πρέπει να υπάρξει λιγότερη παραγωγή. από την άλλη όμως αυτό συνδέεται άμεσα με την άσκηση του επαγγέλματός τους. Ε, εκτός λοιπόν, ε, ή μάλλον σε αντάλλαγμα ε, με την βοήθεια, πρέπει να μειώνεται ο όγκος της παραγωγής που τελικά τίθεται στην αγορά. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι μια ολοκληρωμένη σκέψη, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε. Εδώ και δύο μήνες η Κίνα αγοράζει ε, χοιρινό κρέας ε, και έχουν αυξηθεί οι τιμές κατά 1,30 ε, ευρώ. Τώρα πόσο θα το θα κρατήσει αυτό δεν ξέρουμε γιατί όλα αυτά τα πράγματα ε, είναι πάρα πολύ ευμετάβλητα. Οπότε μας θέσατε έναν προβληματισμό τον οποίο πρέπει να σκεφτούμε Υπάρχει και η γνωμοδότηση της κυρίας Ντολαέ, βεβαίως, όσον αφορά τη διακύμανση των τιμών. 23 Ιουνίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι ε, μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε 1η Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Προπολογισμών. Επίσης ε, 8 Νοεμβρίου θα ψηφίσει ε, η Επιτροπή Γεωργίας και ε, θα εγγραφεί στην Ολομέλεια της, ε, του Δεκεμβρίου. Κύριε Αλή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά έκαναν πολύ πολύτιμα σχόλια. Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, πολύ ευρύ, καλύπτει πολλούς τομείς και ο αγροτικός τομέας δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα ε, ως μεμονωμένος τομέας. Γνωρίζουμε ότι σε παγκόσμια κλίμακα ο γεωργικός τομέας επιδοτείται. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή πολιτική ότι πρέπει να διατηρηθεί η πολιτική αυτή, όμως δεν είναι δυνατόν να προσεγγίζουμε ε, με τον ίδιο τρόπο τον γεωργικό τομέα από καθαρά οικονομική άποψη, γιατί ο τομέας ε, αυτός ε, δεν μπορεί να κριθεί μόνο από τους οικονομικούς δείκτες, η απόδοσή του τουλάχιστον, ε, υπάρχει και το θέμα της ρύθμισης, ε, υπάρχει και το θέμα ε, της φύσης, είναι ένας παράγων εντελώς αστάθμητος που πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Είναι σημαντικό να έχουμε τις απαραίτητες νομές και τους μηχανισμούς για να ρυθμίζονται οι διαδικασίες. Εγώ προσπάθησα να σας παρουσιάσω ε, μια εξισορροπημένη άποψη. Ε, έχουμε λάβει υπόψη και το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Ελπίζουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη έκθεση και θέλουμε όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των συναδέλφων να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πρέπει βέβαια να μπορούν να ε, λένε τις απόψεις τους και οι γεωργοί ε, και να υπάρχει και μια ισορροπία μεταξύ των αγοραστών και των παραγωγών. Είναι σημαντικό να γίνεται αυτό. Όταν ε, οι παραγωγοί πετρελαίου συγκεντρώνονται για να αποφασίσουν ότι θα μειώσουν την παραγωγή ώστε να περάσει το βαρέλι του πετρελαίου από τα 28 στα 25 δολάρια, δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Συνεπώς πρέπει και γεωργοί να ε, συνεταιρίζονται, να ε, ανήκουν σε συλλόγους και να μπορούν να κάνουν το ίδιο, γιατί διαφορετικά θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Η κυρία Γκαρδία Ζαπάλ μπορεί να αντικαταστήσει την κυρία Μούντι όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων από τον προϋπολογισμό Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, ακριβώ όπω είπατε κυρία Μούντι, δεν μπορούσε σήμερα να παραστεί και να μα ε, εξηγήσει τα τη ε, γνωμοδότησή τη. Πρόκειται για κείμενο που απευθύνεται στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Θα την καταρχήσω όσο γίνεται περισσότερο, μια που σε αυτή την έκθεση μιλούμε για την χρηματοδότηση των ε, ΜΚΟ από πλευρά του προπολογισμού. Και η κυρία Μούντι θέλει να το το έργο το οποίο επιτελούν αυτές οι μη οργανώσεις. Να αναγνωριστεί επίσης ότι έχουν έναν ρόλο πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις ευρωπαϊκέ πολιτικές και όχι μόνο στις πολιτικές εκείνε που ε, μπορεί κανεί να του ε, αποδώσει αρμοδιότητα όπως πούμε ανθρωπιστικά αλλά και, αλλού όπως τα πολιτιστικά ε, κλπ. Δηλαδή αναπτύσσουν δραστηριότητα σε πάρα κατευθύνσει και επίσης αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι δεν έχουμε έναν ορισμό νομικό για τα νομικά αυτά προσπαγωμένω. δεν μπορούμε και να υπολογίσουμε τι τμήμα του υπολογισμού θα τους δώσουμε για να πιάσει τόπο. Οπότε αυτό το οποίο προτείνει η συγκέντρια είναι θέλουμε να υπάρξουν κάποια αποτελέσματα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους σχετικούς ε, δείκτες για τα χρήματα του προπολογισμού ανάλογα και βέβαια με το έργο που επιτελούν οι ΜΚΟ. Και αυτό το θέμα επομένως το συζητάμε και το ξανασυζητάμε οι ΜΚΟ αλλά βέβαια και την άλλη μεριά τις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε θέλουμε να είναι πιο άμεση, πιο αποτελεσματική η πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει να λύσει αυτό το πρόβλημα και να βελτιώσει την κατάσταση απλουστεύοντας την. Βέβαια και αυτό αφορά όχι μόνο τον προπολογισμό και τη ΜΚΟ, αλλά και γενικότερα ό,τι χρηματοδοτεί ο που συζητάμε. Επομένω, χρειάζεται να δούμε και τι θα γίνει με το ύψο τη συγχρηματοδότηση. Γιατί έχουμε πάρα πολλέ ΜΚΟ, οπότε πολλέ φορέ είναι τόσο υψηλή η χρηματοδότηση που εμποδίζει τη συμμετοχή των ΜΚΟ στα έργα και προγράμματα. Άρα θα πρέπει και αυτό να μελετηθεί και θα πρέπει τελικά ε, ο πύχης να μην πηγαίνει παραπάνω από το 20%. Ε, επίσης όσον αφορά την συγχρηματοδότηση αναφέρεται και κάτι άλλο. Θα πρέπει βέβαια αυτό να το συνοηθούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας πει τι συμβαίνει. Θα πρέπει επομένως να εμβαθύνουμε και να δούμε τι μπορούμε να καταλογίσουμε στην συγχρηματοδότηση. Ε, γιατί έχουμε και κάποιους φορείς ε, εθελοντικής φύσεως μέσω αυτών. Επίσης, ε, όσον αφορά την απορροφητικότητα και απορρόφηση των πόρων, ισχύει το use it or lose it. Πολλές φορές δηλαδή θα πρέπει για να μην χαθούν οι πόροι να βιαστούν αυτά τα νομικά πρόσωπα, να τους ε, ε, αξιοποιήσουν. Και αυτό βέβαια δημιουργεί ζητήματα όσον αφορά το κατά πόσον οι πόροι πιάνουν τόπο. Έχουμε κάποιους τροπολογίες ε, πολλές που έχουν υποβληθεί από ό,τι μου λέει η κυρία Μούντι πολλές από τις τροπολογίες μπορεί να αγκαλιάσει η έκθεση μπορεί να γίνουν και συμβαστικές τροπολογίες θα τα πούμε τις επόμενες μέρες Ευχαριστώ κύριε Καλίστα Η κυρία Φάνα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μούντι για την γραμμοδότησή της σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Τον έλεγχο τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό το θέμα αυτό, γιατί όπω είπε η συνάδελφο, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο αντίκτυπο τη εργασία των ΜΚΟ και δεν περιορίζεται μονάχα στην σημασία που έχουν για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μονάχα η επιρρογνωμοσύνη που δίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά βοηθούν στην πράξη να εκτελεστούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ευρώπη 2020 και μας επιτρέπουν να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει λοιπόν να παραγνωρίζεται ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να θεωρείται ότι είναι ένα δευτερεύον περιθωριακό θέμα. Η γνωμοδότηση είναι μια καλή γνωμοδότηση, μια πολύ καλή βάση συζήτηση, όπως είπε και η κυρία Γουάρια Σαβάλ, αφορά περισσότερο τις μικρότερες ΜΚΟ που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες και έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος. και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι γέννη μια απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους, ιδίως τουλάχιστον στη φάση που θα πρέπει να εκτελεστούν τα προγράμματα και να ελέγχονται οι πιστώσεις οι οποίε δίνονται. Εμεί έχουμε καταθέσει ορισμένε τροπολογίες με στόχο να απεικονίσουμε καλύτερα την ε, δραστηριότητα των ΜΚΟ και τον ρόλο τους για την πραγματικότητα. Παραδείγματος το, η οροφή για τα έμεσα, για το έμεσο κόστος από το 7% θα πρέπει να ανέλθει στο 15%. Έχουμε μια τέτοια τροπολογία. Αυτό περιλαμβάνεται σε μια α, ρήτρα εξαίρεσης η οποία απαιτεί μια γνωμοδότηση θετική της Κομισιόν. Εδώ όμως μπορεί να αυξηθεί αυτό το ε, όριο γιατί υπάρχουν προγράμματα του, της Ευρώπης 2020 που έχουν έμεσο κόστος το οποίο φτάνει το 25% του συνόλου. Μπορούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε μικρομεσαίε επιχειρήσει και επίση να έχουμε και ένα μηχανισμό επίλυση διαφορών που θα δίνει δυνατότητα στι ΜΚΟ σε περιπτώσει που υπάρχει μια διαφορά με την Κομισιόν να επεμβαίνει κάποιο διαμεσολαβητή και να βρίσκει μια κοινή αποδοχή λύση. Αυτό μέχρι στιγμή δεν έχει επιτευχθεί Εν κατακλείδη θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή η γνωμοδότηση, αλλά πιστεύω ότι πάντα μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω και εμείς θέλουμε να τονίσουμε την ε, απλοποίηση και τη μείωση του άκτους για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία Κυρία Σουλίν. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Σουλίν. Και εγώ μπορώ να συμφωνήσω με τους ε, προλαλήσαντες και τις προλαλήσασες. Είναι πολύ σημαντικές οι ως στην κοινωνία. Εκπληρούν κάποιους ρόλους που δεν μπορούν να τους καλύψουν οι κυβερνητικές οργανώσεις. Και στα πλαίσια της τωρινής κρίσης μετανάστευσης, με την μεγάλη ροή προσφύγων, είδαμε να υπάρχει όλο και μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των ΜΚΟ στις χώρες μας και ιδίως στα κέντρα υποδοχής προσφύγων. Εδώ μας ενδιαφέρει το θέμα του ελέγχου της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συγγνώμη, των ε, σε αυτές τις ενέργειες. Κάποιοι έλεγχοι μας οδηγούν στο να κατανοήσουμε ότι χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα η ΜΚΟ για δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να είναι και αντιευρωπαϊκές. Και αυτό φυσικά δεν συνάδει με τις κέρυες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν οργανώσεις που χρησιμοποιούν τα κονδύλια μας για ρατσιστικούς, αντισημιτιστικούς και άλλους συναφείς σκοπούς. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει στην ε, λειτουργία <clears throat> της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη πολλές φορές σε ορισμένες ΜΚΟ χρηματοδοτούν άλλες ΜΚΟ. Αυτός όμως είναι αδιαφανής τρόπος για να χρηματοδοτείται το έργο των ΜΚΟ από το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να χρηματοδοτήσει μια συγκεκριμένη ΜΚΟ, αλλά έμεσα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περαιτέρω ελέγχους και περαιτέρω αξιολογήσεις για τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Πρέπει να ελέγξουμε και να εξασφαλίσουμε τα προγράμματα που εκτελούν οι ΜΚΟ έχουν σαφώς καθορισμένους στόχους και οι στόχοι αυτοί συνάδουν με τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ΜΚΟ και σε περίπτωση καταχρήσεων και παραβιάσεων, θα πρέπει να ζητήσουμε τα χρήματα αυτά όσον να επανέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εάν αυτό είναι απαραίτητο, μια ΜΚΟ η οποία έχει ε, καταχρηστεί των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων θα πρέπει να υποστεί και κυρώσει. Όταν γίνεται παραδείγματο χάρη πρόσκληση ενδιαφέροντο για νέα σχέδια, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυτέ οι ΜΚΟ. Κύριο Μπόκετ. Μπόκετ, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην πραγματικότητα, πολλές ΜΚΟ διαδραματίζουν μια εξαιρετικά σημαντική εργασία στην, ε, στην κοινωνία μας. Αλλά πρέπει να δώσω και δίκιο στην προλαλήσατα. Πολλές φορές γίνεται μια αδιαφανής χρησιμοποίηση των κονδυλίων για σκοπούς οι οποίοι δεν είναι απαραίτητοι. Το έχουμε δει ήδη στο παρελθόν ότι πολλές φορές με ε, ένα είδος προπαγάνδας και μισοαληθιών γίνονται κάποιες, ε, ε, δημιουργούνται κάποιες εντυπώσεις οι οποίες δεν προωθούν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι λέγονται πράγματα τα οποία παραπλανούν τους πολίτες για τα θέματα της ανάπτυξης. Νομίζω ότι το να υπάρχουν μηχανισμοί για την διαμεσολάβηση, ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να προχωρήσουμε περισσότερο για να επιλύουμε τέτοιες διαφορές. Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ένα θέμα που αντιμετωπίσαμε στην Επιτροπή ΙΝΤΑ για τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές ενέργειες πάντα υπήρχε μια συμφωνία ότι πρέπει να υπάρχει και κάποια έκθεση ε, που να προβλέπει τι θα προέλθει από ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα. Αλλά εγώ πρέπει να διαπιστώσω ότι υπήρξε μια μελέτη από την Κομισιόν για το ρόλο του ΜΚΟ σε ό,τι αφορά τις ε, συμφωνίες εξωτερικού εμπορίου. Αυτό όμως το κείμενο έχει αποσυρθεί. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι το οποίο είχαμε συμφωνήσει να γίνεται από την Κομισιόν να μας παρουσιάζει τέτοιου είδου κείμενα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω και από τους συναδέλφους της Κομισιόν που ήταν παρόντες στην Επιτροπή Ίντα και οι οποίοι προσπάθησαν να βγάλουν την ουρά τους και να αποσύσουν την ε, ευθύνη τους να φέρουν σε πέρα στο έργο τους έναντι του Κοινοβουλίου γιατί ξέρουμε ότι από αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού έχουν εκτελεστεί ε, μελέτες, επομένως υπόκειται η Κομισιόν στην υποχρέωση να μας παρουσιάζει μια ανακοίνωση, μια ε, ανακοίνωση μέχρι το καλοκαίρι για το τι θα κάνει με αυτές τις διαδικασίε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κομισιόν να συνεχίζει τη χρήση αυτή τη γραμμή του προπολογισμού χωρίς να μας δίνει ε, εκθέσει για τα θέματα αυτά. Αν η Κομισιόν λοιπόν ακολουθήσει μια στάση άρνηση, θα πρέπει εμείς να κάνουμε τι απαραίτητε αλλαγέ στον προπολογισμό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο, την ε, κυρία ε, Μούντι και ως θα ήθελα να πω ότι 32 τροπολογίες έχουν κατατεθεί και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο τις καταθέσατε. Ο κύριος Νεγκρέσκου έχει καταθέσει την ε, πλειονότητα των τροπολογιών αυτών, αλλά συμφωνούν όλες ε, με την θέση του ΕΛΚ και πιστεύω ότι τις περισσότερες θα τις υποστηρίξω. Θα ήθελα τώρα να πω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις κατά την άποψή μου, επιτελούν έργο πάρα πολύ καλό, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις αντίθετες. Και ε, επειδή κάποιες από αυτές τις οργανώσεις δεν ε, επιτελούν σωστό έργο, δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε όλα αυτά που αναφέρθηκαν σε αυτήν την έκθεση. Στη γνωμοδότηση αυτή πρέπει να αναφέρεται σαφέστατα ότι θέλουμε διαφάνεια, να ξέρουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα και ότι αν εγκρίνουμε τις τροπολογίες και την ίδια την έκθεση, η οποία είναι πάρα πολύ καλογραμμένη, πρέπει να το πω αυτό, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, στον ε, κόσμο των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, σαφώς υπάρχει τεράστια ποικιλία. Μπορεί να συμβεί το ότι η διενέργεια περισσότερων ελέγχων ε, μπορεί τελικά να γίνει κάτι το εντελώς μη βιώσιμο. Ε, στο Λίβανο και στην ε, Ιορδανία είδαμε κόσμο για παράδειγμα της UNICEF που ήταν αντικείμενο ελέγχου, ελέγχων, 10 ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μία χρονιά. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε κάπως να συντονίσουμε αυτούς τους ελέγχους ενδεχομένως και να τους αποφύγουμε. Αυτή τη στιγμή βέβαια εξασφαλίζεται η διαφάνεια και ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε σχέση με το πού προέρχονται οι, ε, οι πόροι. Μερικές φορές ε, είναι τα πράγματα πολύ ομιχλώδη και αυτό δεν μπορεί να ε, συνεχιστεί. Η εμπιστοσύνη προέρχεται από τη διαφάνεια, αυτό είναι βέβαιο. Ίσως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να απαντήσει στον κύριο Μπέγκε. Ε, Euh, Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ε, θα ενημερωθώ και αν θέλετε διμερώς ε, ευχαρίστως να σας ε, παράσχω όλα τα στοιχεία. Θα ήθελα να κάνω όμως μερικά σχόλια, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την ε, συζήτηση, η οποία είναι ε, πάρα πολύ πλούσια, και να αναφερθώ σε μερικά ζητήματα που αναφέρθηκαν. Καταρχάς, πράγματι η προσπάθεια απλοποίησης και εναρμόνισης ε, είναι στόχος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως επικροτούμε την, το σχέδιο γνωμοδότησης ε, ως προς αυτό. Όσον αφορά το θέμα της συγχρηματοδότησης, ε, μέγιστη συγχρηματοδότηση και αν θα έπρεπε να εφαρμοστεί αυτή ο ε, κανονισμός ο δημοσιονομικός δεν προβλέπει συγκεκριμένο επίπεδο. Σε, κάποιο, σε κάποια τομεακή βάση μπορεί να υπάρχει ένα μέγιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης το οποίο να δεσπίζεται για συγκεκριμένους στόχους ε, πολιτικών ε, στο πλαίσιο χρηματοδότησης ενός προγράμματος, αλλά νομίζω ότι όταν αποφασίζουμε ποιο είναι το βέλτιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης πρέπει να εξετάζουμε όχι μόνο την λειτουργία ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο ε, των ε, ενωσιακών κονδυλίων με, σε σχέση με το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε και ένα πολύ ψηλό ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να δημιουργήσει και μια σχέση εξάρτησης, ε, κάτι το οποίο μπορεί να ε, δημιουργήσει πρόβλημα και μπορεί να δημιουργήσει μετά και πρόβλημα στο να λάβουν τέτοιου είδους κονδύλια και νέο εισερχόμενοι στο πρόγραμμα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία που να επιτρέπει να μεγιστοποιεί το αντίκτυπο, να μεγιστοποιείται το αντίκτυπο, ο αντίκτυπος όλης αυτής της διαδικασίας. Θα ήθελε επίσης να πω ότι η εισφορά σε είδος δεν είναι δυνατόν ε, να ε, αμείβεται με κάποιο τρόπο συγχρηματοδότησης που προκύπτει από τον ίδιο το μη κυβερνητικό οργανισμό. Ε, είναι γεγονός ότι το τέτοιου είδους ε, ε, συνεισφορά συνήθως, σε είδος δηλαδή συνεισφορά, συνήθως ε, λαμβάνεται υπόψη στο σύνολο της χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Καρδιαζαμπάλ, για να συνοψίσει εκ μέρου της κυρίας Κούντι. Ναι, είναι περίπλοκο αυτό να συμφωνήσουμε γιατί θα διαβιβάσω αυτά τα οποία προτείνεται στην κυρία Μούντις και επίσης θα τις διαβιβάσω της Παρτίδης Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Να σας πω κάτι, κάτι που είναι δικό μου Αυτό όσον αφορά το τι μετράει η φροντική εργασία, πρόσφατα πρόσφαση σε είδος, γιατί ε, έχουμε αντιμετωπίσει και πάλι το πρόβλημα αυτό και πολλές μη και όχι και κάποιες οργανώσεις ε, των νεολαίων λένε το αντίθετο, οπότε είναι δύσκολο κανείς να καταλήξει σε κάποια τοποθέτηση. Πάντως, εγώ θα τα πω όλα τα σχετικά στην κυρία Μούντι, θα κάνει αυτές τις προτάσεις της για συμβαστικές τροπολογίες και θα πάμε μετά για την ψήφιση. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα είναι επομένως ε, αυτό στις 23 Ιουνίου και πιο μετά θα είναι στις 30. Ευχαριστούμε κύριε Κατία 30 Σύρια πρόσφυγες Παλαιστίνιου, πολλοί εκ των οποίων πήγανε σε Ιορδανία και Λίβανο άρα σκεφτείτε τι περάνθρωπες προσπάθειες έπρεπε να καταβάλουν αυτές οι δύο χώρες ούτως ώστε να αναδεχθούν αυτούς τους ε, πρόσφυγες με τόσο πολύ βλέπετε επομένω ότι παρενέβη χρηματοδοτικά η Ευρώπη και αυτό ε, ήταν αυτοί οι οποίοι υπηρετούν στις ε, αντιπροσωπείες της Ένωσης με επαγγελματικό τρόπο και παραβάλλουν μεγάλες και χρειάζεται ενίσχυση επομένως από σχεδόν δεν τα δικαιούνται επισήμως τότε έχουν πρόσφυγες από τη Συρία είναι ότι περιμένανε να επανέλθει η ειρήνη στη Συρία για να μπορέσουν να γυρίσουν στις αιστείες τους και θα πρέπει να ασκήσει πίεση η Ευρώπη για την επαναφορά της ειρήνης στη Συρία. Το έγγραφο αυτό λοιπόν σας έχει διανεμηθεί, ελπίζω να το διαβάσετε και στρέφομαι κυρίως προς τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετέσχαν σε αυτή την αποστολή θα ήταν χρήσιμο αν μπορείτε να μου δώσετε και τα σχόλιά σας πριν από την Τετάρτη 22 Ιουνίου για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε αυτό το κείμενο. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της Κομισιόν για την αρρωγή που μας έδωσαν. Ιδίω αυτούς που ήταν επιτόπου στις χώρες που επισκεφτήκαμε ήταν πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. και τον κύριο Μουράκη κυρίω και τον Κάσιο Αμαλέ που μας βοήθησαν πάρα πολύ στο έργο μας επιτοπίως για να γίνει καλά η εξέλιξη αυτής της αποστολής που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Σύσταχουν τώρα στους συναδελφούς που ήταν μέλη της αποστολής αν έχουν να κάνουν κάποια σχόλια, θέλουν να προσθέσουν κάτι σε αυτά τα οποία είπα. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Α, κύριε Γκάιερ. Εγώ δεν μπόρεσα να λάβω μέρος σε αυτή την ε, αποστολή, αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτά που αναφέρατε, τα κριτικά σημεία τα αναφέρατε, μου θυμίσουν την εποχή που εγώ ήμουνα σε, ως ε, στην ε, Βόρεια Ιρλανδία Βεσφαλία σε μια εταιρεία περιορισμένη ευθύνη. Εκεί υπάρχουν δύο μορφές επικρίσεως που μπορεί κανείς να, διατυπώσει για επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν με δημόσιο χρήμα. Πάνω σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία εργαζόμενα, συγγνώμη. Αν τηρήσει κανείς όλους τους κανόνες που έχει, τότε τα πράγματα προχωρούσαν με ρυθμό χελώνα. Αν... Και αν δεν τηρήσει κανείς τους κανόνες, τότε είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Του λέγανε ότι εάν κάνεις κάποιο λάθος, τότε πώς εσύ έκανες μια τέτοια διασπατάληση δημοσίου χρήματος το οποίο σου δίνει ο φορολογούμενος, ο Γερμανός ή ακόμα και ο Ευρωπαίος. Η Κομισιόν σίγουρα έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλία για κάποιο έλεγχο γιατί πολλά πράγματα είχαν γίνει χωρίς, ε, χωρίς έλεγχο. Πάντα οι έρχονται αυτοί από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και λένε ε, επί τη βάση και ορισμένων εκθέσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου, έχουν επικρίνει την Κομισιόν γιατί δεν έκανε τους απαραίτητους, κατά την άποψή τους, ε, ελέγχους και ζητούν πάντα μία αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων. Τότε γίνονται αυτοί πιο <clears throat> ενδελεχείς ε, έλεγχοι και βλέπουμε στην, την επίπτωση που έχουν, το είδαμε αυτό στη Μέση Ανατολή, οι φορείς αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν σε πίεση από την Κομισιόν ότι είναι υποχρεωμένοι να προχωρούν πολύ αργά λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων. Επομένως, η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη τη μια φορά να λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να λειτουργήσει πιο γρήγορα, άλλη φορά να λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να έχει πιο αυστηρούς ελέγχους, αλλά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να σκεφτεί λιγάκι καλύτερα για το θέμα αυτό. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει κάποια λύση, αλλά θέλω εδώ να πω ότι δεν φταίει και η Κομισιόν, γιατί ό,τι και να κάνει θα είναι παράπτωμα. Θα την επικρίνουν ή για τη βραδύτητα ή για την έλλειψη ελέγχων. Εγώ δεν θέλω να γίνουν τα πράγματα εκτός ελέγχου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι στο Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό ελεκτικό ε, συνέδριο που θεωρούν ότι αν δίνει χρήματα σε κάποιο καταπίστευμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στα Ηνωμένα Έθνη, στην UNICEF που τα χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα του καταστε... καταπιστεύματος για να φτιάξουν σχολεία, θα πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά μέχρι και το τελευταίο τούβλο. Τα λέω λιγάκι χοντρά. Αλλά όταν πρόκειται για την χρηματοδότηση, Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι λίγο πιο εξισορροπημένο στην κριτική που ασκεί στην Κομισιόν, να υπάρχει μόνο το επίπεδο ελέγχου που είναι απαραίτητο και να υπάρχει η απαραίτητη ευκαμψία στην Κομισιόν και ίσως μπορούμε να είμαστε λιγότερο επικριτικοί κατά της Κομισιόν αλλά πάντα είναι πολύ δύσκολο να βρει κανεί τη σωστή ισορροπία, γιατί για ορισμένου είναι πολύ γραφειοκρατική, για άλλου είναι πολύ χαλαρή. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε και στο πλαίσιο της πολιτικής που χρηματοδοτούμε. Το κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε τους πολιτικούς στόχους και όχι μονάχα τους στόχους ελέγχου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να ελέγχουμε για την καλή χρησιμοποίηση των δημοσίων κονδυλίων, αλλά ο υπερβολικός έλεγχος σκοτώνει τον έλεγχο. Μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που τελικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Σήμερα το πρωί <clears throat> ανέφερα μία εμπειρία που έζησε με ένα πιλωτικό σχέδιο για τα, το χαρτοβασίλειο που ζητάει η Κομισιόν για να δώσει 5 ευρώ. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν είναι πια λογικό. Δεν είναι μονάχα το θέμα του ελέγχου, αλλά θα πρέπει να δούμε την ουσία του προβλήματος και όχι σε μια κατάσταση κρίσης να ζητάμε από τους ε, πυροσβέστες να κάνουν εξοικονόμηση νερού όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν πυρκαγιές. Οι αρχές του Λιβάνου και μας το είπανε και συναντήσαμε και υπουργούς και βουλευτές Θέλουμε, τους είπαμε, η κυβέρνηση να παρουσιάζει λογαριασμούς οι οποίοι να είναι διαφανείς. Και εκεί έχουμε να κάνουμε, ακόμα κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει να αναφερθεί στην έκθεση πεπραγμένο στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Αλλιώ πηγαίνουμε στι ψηφοφορίε. Κύριε Μαραγκάλ, θέλετε να πείτε κάτι. Μόνο θα ήθελα να πω εξ ονόματο τη Μόνικα Βάνα που χρειάστηκε να φύγει να κάνω δύο πάρα πολύ σύντομες ε, παρατηρήσεις έχοντας στο μυαλό μου την ε, μνήμη της προηγούμενης επίσκεψής μας στην ε, Τουρκία που είχε κάποιες διαφορές με αυτά που είδαμε στην, που αναφέρατε για την Ιορδανία και το Λίβανο. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η κατάσταση στο Λίβανο και την η Ορδανία δεν είναι καλύτερη, αλλά είναι μάλλον χειρότερη σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και χρειάζονται να υπάρχουν ειδικέ πολιτικές για τους πρόσφυγες εκεί, ιδίω για αυτούς που είναι σε επισφαλή κατάσταση. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι τα κονδύλια που πηγαίνουν προς τους πρόσφυγες θα πρέπει να λαμβάνουν και την κατάσταση της κοινότητας όπου ζουν οι πρόσφυγες δεν πρέπει να είναι χρήματα που δίνονται μονάχα στους ε, πρόσφυγες, αλλά και στην ε, κοινότητα που τους υποδέχεται για τη βελτίωση των βασικών υπηρεσιών, της υδροδότησης, της ε, υγειονομικής περίθαλψης κτλ. Και επίσης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα που έχουν σαν στόχο να υποστηρίξουν την πολιτική ισότητα των φύλων γιατί αλλιώς έχουμε δει να υπάρχουν απαράδεκτες καταστάσεις άσκησης βίας, ιδίως σεξουαλικής βίας για έναντι των γυναικών που είναι πρόσφυγες και η Μόνικα Βάνα μου ζήτησε να υπογραμμίσω ιδιαίτερα αυτές τις πτυχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρος. Εγώ δεν είπα απλώς για τους ίδιους πρόσφυγες που είναι στα σύνορα της Ιορδανίας, είναι κάπου 50.000 οι οποίες βρίσκονται σε πάρα πολύ άθλιες συνθήκες. Μετά από την επίσκεψη του πρόεδρου Ομπάμα, δέχτηκαν οι Ορδανοί να δέχονται κάθε μέρα 200-300 πρόσφυγες. Αυτό βέβαια δεν λύει το πρόβλημα των υπόλοιπων. Πράγματι όμως ως Ευρωπαίοι δεν θέλουμε, δεν δίνουμε καλύτερες συνθήκες υποδοχή των προσφύγων εδώ στην Ευρώπη από αυτά που γίνονται στην ε, περιοχή κοντά στη Συρία. Σκέφτομαι με χάρη τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο Καλέ και θέλουν να πάνε στη Μεγάλη Βρετανία και δεν μπορούν να πάρουν να το κάνω αυτό. Λοιπόν, τα σχόλιά σας μέχρι τις 22 του μηνός για να κλείσει αυτό το θέμα. Ψ, ψηφοφορίες τώρα παρακαλώ βάλτε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες στο αντίστοιχο σύστημα και να κάνουμε μια πρώτη προσωμείωση ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Προσπαθώ να δω ποιος είναι ο αριθμός των ψηφισάντων. Κάποιος από εσάς δεν ψήφισε. Τώρα. Πέρας. Έκθεση Φερνάντες. Διορθωτικός προϋπολογισμός υπερθυμών 2, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία επαγγελμών 4. Πέρασε. απορρίπτεται. 8-16 απορρίπτεται. Τροπολογία 5 απορρίφθηκε, ε, αποσύρθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9, 10 και 11 θεωρούνται μη παραδεκτές. Το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση παρακαλώ, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται ο διορθωτικός προπολογισμό με 25 ψήφους υπέρ εναντίον μίας και με μία αποχή. Έκθεση του κυρίου Νεγκρέσκου για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία 2. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 εκπίπτει. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 11 υπέρ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 14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 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 22. Το πρώτο τμήμα της έχει εκπέσει λόγω της έγκρισης της τροπολογίας 21 και ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα το οποίο είναι συμβατό με την ε, τροπολογία 21. Δεύτερο τμήμα της 22. Συμβατό με την 21. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Θα ελέγξουμε για την 23. Πέρας. Εγκρίνεται. 13-11. 24 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16-10. 25 εκπίπτει διότι είναι κρίτη 24, 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται το σύνολο του κειμένου. Όπως έχει τροποποιηθεί άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ενεκρίθη. 24 εναντίον τριών. Ο κύριος Φερνάντες για τις ε, μεταφορές πιστώσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα παρουσιάσω ξεχωριστά, που θα τα ψηφίσουμε ξεχωριστά. Για τη μεταφορά 8 1.824.042 ευρώ για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για το Βέλγιο ε, και θα ήθελα να ψηφίσουμε υπέρ. Δεύτερο, ε, δεύτερη μεταφορά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει λίγο περισσότερα πράγματα για αυτό το έμβασμα. 50 εκατομμύρια για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διασύνδεσης στην Ευρώπη για τις τηλεπικοινωνίες εν ώψη της ε, δημιουργίας ενός ε, νέου δικτύου υψηλ... ευρυζωνικού δικτύου. Ε, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα σε σχέση με αυτό το νέο ε, μέσο όπως επίσης και το ρυθμό εφαρμογής ε, του Connecting Europe ε, Facility και την πτυχή της ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά. Η ιδέα όσον αφορά την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη είναι να επισπεύσουμε ε, την επικοινωνία και την τεχνολογία και να πρικοδοτήσουμε εγκαίρως ε, τις δράσεις που αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Η ιδέα είναι να, δημιουργήσει ένα, να δημιουργηθεί ένα επενδυτικό ταμείο για, την, ε, για το ευρυζωνικό δίκτυο που σημαίνει υψηλής ταχύτητας ευρεία ζώνη ε, και η εστίαση θα αφορούσε μικρότερης κλίμακας αλλά υψηλού κινδύνου ε, έργα, ώστε με ε, οι υποχρεώσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα συμμετοχής και άλλων παικτών της αγοράς και όπως και επίσης συλλογή πιστώσεων 450 εκατομμυρίων, 400 από τον υπολογισμό και τα 50 εκατομμύρια τα επιπλέον για τα οποία μιλούμε θα μας δώσουν τη δυνατότητα το 2016 να συγκεντρώσουμε όλο το ποσό. 100 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναμένονται περίπου 100 με 120 εκατομμύρια από εθνικές τράπεζες ε, προώθησης ε, ε, και ε, 100 ε, με 120 εκατομμύρια είναι το ποσό που αναμένεται αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει αλλαγή όσον αφορά την, το, το κομμάτι της διευκόλυνσης που πηγαίνει στην ενέργεια. Απλώς γίνεται μία μεταφορά ε, με προχρηματοδότηση, αύξηση της προχρηματοδότησης που αφορά το κομμάτι για το Ευρυζωνικό Επενδυτικό Ταμείο ε, και η ενεργειακή πτυγή θα καθυστερήσει και θα αντισταθμιστεί το 2018. Επομένως το ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό δεν τροποποιείται και στην περίπτωση της ενέργειας ε, το 2016 κάποια από τα προγράμματα ε, τα οποία παρουσιάστηκαν ε, στην προκήρυξη του διαγωνισμού δεν θεωρήθηκαν ότι ήταν αρκετά όρημα για χρηματοδότηση. Κάποια από τα στοιχεία δεν ε, πληρούσαν τα απαραίτητα οικονομικά, τις απαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμα. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το κομμάτι της ε, τεχνολογίας, της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε όσον αφορά τις ευρυζωνικές δραστηριότητες, ενώ η ενεργειακή πτυχή, η ενεργειακή επένδυση θα καθυστερήσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστω να απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ισηγητά, μήπως οι πληροφορίες αυτές είναι επαρκείς ε, και ενισχύουν την άποψή σας ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε. Ναι, εγώ όμως το ερώτημα το έθεσα, για να, το ρώτησα για να είναι η Επιτροπή μας ε, καλύτερα ενημερωμένη. Πιστεύετε ότι μπορείτε να ψηφίσετε λοιπόν πιο ενημερωμένα. Ωραία, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. 22 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και δύο αποχές. Μικρόφωνο παρακαλώ. Πολύς μικρόφωνο κύριε Στεπρέ. 3.126 περίπου ευρώ για την Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Σχολείο της Φραγκφούρτης. Αυτό λόγω της καθυστέρησης των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ΙΟΠΑ για την χρηματοδότηση αυτού του σχολείου, του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Θα ήθελα να ξέρω και ίσως η Κομισιόν μπορεί να μας το εξηγήσει εδώ ποιες ακριβώς ήταν οι δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν σε αυτή τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με την ΙΟΠΑ και κατά πόσο θα επιληθούν ταχαίως ή όχι. Με αρνητικά επιτόκια βέβαια η Κεντρική Τράπεζα, λέει ο πρόεδρος, έχει αρκετά λεφτά στο Ευρωφυλάκειό της. Παρακαλώ κύριε Φρέζα. Σας ευχαριστώ. Να σας εξηγήσω στην αρχή πώς λειτουργούσε στον προϋπολογισμό η δαπάνη για τα ευρωπαϊκά σχολεία και ιδίως στην περίπτωση φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και έχουν το δικό τους αυτόνομο προϋπολογισμό με την αύξηση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυξήθηκε και ο αριθμός των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο στη Φραγκφούρτη και τώρα έχουμε μια μεγαλύτερη διοικητική δαπάνη η οποία βρίσκεται στον προϋπολογισμό της Κομισιόν. Γιατί τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι στον προϋπολογισμό της Κομισιόν. Και τα σχολεία αυτά φυσικά δεν έχουν να κάνουν με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, αλλά εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής ε, Κομισιόν. Της Κομισιόν. Προσπάθησε λοιπόν η Κομισιόν να πει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλους φόρους, άλλους φορείς που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά σχολεία ότι πρέπει να υπάρχει μια δίκαια καταναμή πόρων για να υπάρξει και διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον καταλογισμό του κόστου των σχολείων να ξέρουμε από πού προέρχεται το κόστος και πού πρέπει να αναφέρεται στον προϋπολογισμό. Εφόσον εδώ πέρα πρόκειται για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα πρέπει να υπάρξει η κατανομή του κόστους και στην Κεντρική <clears throat> Τράπεζα, η οποία έτσι θα συνέβαλε στην σχολική εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού τους. Οι διαπραγματεύσεις ε, είναι σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες δεν υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός για να αλλάξουν οι συμφωνίες για τη χρηματοδότηση, αλλά υπάρχει πρόοδος. Υπάρχουν άλλοι φορείς ε, όπως το Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπου υπάρχει ένα αντίστοιχο καθεστώς και έχουν οδηγήσει σε κάποια συμφωνία αυτέ οι συμφωνίε. Για το 2016 όμω η Κομισιόν δεν ήταν σίγουρη ότι θα μπορούσε να περατωθεί εν αυτή η διαπραγμάτευση και γι' αυτό πρότεινε να εγγραφεί το αντίστοιχο ποσό στο αποθεματικό για να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δεχόταν να δώσει τη συμφορά της εγκαίρωσης. Ο δημοσιονομικός κανονισμός τώρα που αφορά τα ευρωπαϊκά σχολεία προβλέπει ότι το 10, τα δέκατα των δαπανών θα πρέπει να είναι διαθέσιμο μέχρι τις 15 Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δώσει τώρα τίποτα. 40% είναι το ποσό που βρίσκεται στο απαθηματικό και γι' αυτό η Κομισιόν παρουσιάζει αυτή την αίτηση μεταφοράς που θα επιτρέψει στο σχολείο της Φραγκούρτης να τηρήσει αυτή την υποχρέωση που έχει μέχρι 15 Ιουλίου. Ο στόχος είναι βέβαια να αντιμετωπιστεί μια μεταβατική κατάσταση γιατί ελπίζουμε από το 2017 θα μπορέσει να υπάρξει η σωστή ο σωστό επιμερισμός κόστους που να περιλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ κύριε Γενική Εισηγητά, είσαστε ικανοποιημένος από αυτά. Χωρίς μικρόφωνο κύριος Φερνάντης. Πιστεύω ότι μπορώ να προτείνω μια θετική ψήφο και για τα διάφορα κύριε Πρόεδρε θα θέσω ένα άλλο θέμα για μια άλλη μεταφορά πιστώσεων για τις αυτόνομες αυτές μεταφορές της Κομισιόν. Και εγώ έχω ένα ερώτημα πριν από την ε, ψηφοφορία, κύριε Φρέζα. Στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βλέπουμε να, έχουν, να υπάρχουν κάποια έσοδα. Αυτά τα έσοδα λοιπόν θα καταλογιστούν αμέσως στις δαπάνες για το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Ναι, δεν έχουμε έσοδα αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην περίπτωση που όταν υπάρχουν έσοδα τότε θα μειωθεί η γραμμή του προπολογισμού από την πλευρά της Κομισιόν. Επομένως αυτό που εμφανίζεται στον προπολογισμό είναι το καθαρό ποσό. Αφαιρούμε τα έσοδα, αλλά δεν δείχνουμε ότι υπάρχουν έσοδα. Απλώς αυτό αφαιρείται από τις δαπάνες. Είναι μια ιδιαίτερη τεχνική αυτό. Ναι, αλλά εμεί εγγράφουμε στον προπολογισμό μονάχα το καθαρό ποσό το οποίο ενδιαφέρει τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και είναι μονάχα η διαφορά μεταξύ της του κόστου και της συνεισφοράς της Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά στο συνοδευτικό έγγραφο υπάρχει η καταγραφή του πλήρους κόστους και αυτό για τους στόχους της διαφάνειας. Υπάρχει πλήρης πληροφόρηση. Εντάξει, ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. <coughs> <coughs> Κάποιος δεν έχει ψηφίσει. Πέρασε. 21-2 γίνεται δεκτή η πρόταση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισηγητά. Κύριε Ντεπρέ, έχετε εσείς κάποιες ε, μεταφορές να προτείνετε. Ναι κύριε Πρόεδρε, τρεις μεταφορές. Η πρώτη αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 1.800.000 από τη θέση 1.200 που αφορά μισθούς και άλλες αποδοχές επειδή ένας αριθμός 7 ε, από τις 12 δικαστές έχουν μπει στη, έχουν αναλάβει τα καθήκοντά τους το 12 που πρόκειται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και υπάρχει επίσης και το θέμα των γνωσικών υπηρεσιών λόγω και της αύξησης του κόστους μετάφρασης τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και προβλέπει το 2017 να μεταφραστούν 53.000 σελίδες παραπάνω από ότι το 2016. Υποστηρίζω λοιπόν αυτή την μεταφορά. Δεύτερη αφορά την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ευρώ από την διερμηνία σε άλλες θέσεις το 2017 για να υπάρξουν μετρητές ενέργειας και να αντικατασταθεί η ηλεκτρική θέρμανση με την ε, θέρμανση με φυσικό αέριο, το οποίο μου φαίνεται οικονομικά λογικό και περιβαλλοντικά λογικό. Και επίσης 6.000 ε, 2.620 για για ε, βελτίωση της αποχέτευσης του κτίριου. Έχω να θέσω για το τρίτο. Θα ήθελα να ψηφίσουμε τα δύο πρώτα, γιατί για το τρίτο έχω κάποια ερωτήματα. Για τα πρώτα δεν υπάρχει καμία ανάγκη ψηφοφορία εκτός αν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Ναι, νομίζω ότι είναι εντάξει. Κύριε Μάνκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. να εκφράσω τη γνώμη για αυτές τις μεταφορές. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι καλό να εξοικονομεί χρήματα και να χρησιμοποιηθούν αυτά οι, αθήποροι για άλλους στόχους, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι χρειάζεται παροχή από υπηρεσιών από εξωτερικούς παροχούς, δηλαδή γίνεται μετάφραση μέσω του ίντερνετ από εξωτερικό προσωπικό είχε πει ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το ε, μόνιμο προσωπικό του και τώρα θέλουμε περισσότερους εξωτερικούς μεταφραστές. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα. Αυτό για μένα είναι σημαντικό ερώτημα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει Κατά υποστηρίζω αυτή τη μεταφορά και δεύτερον για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εντάξει, 400.000 εξοικονόμηση για την διερμηνία, θα μειωθεί και η κατανάλωση ενέργειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δεχόμαστε. Αλλά και εδώ πρέπει να πω το εξή. Θα γίνουν εξοικονομήσεις στη διερμηνία, αλλά χρειαζόμαστε και περισσότερες πληροφορίες. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι θετικό και για τους διερμηνείς. και αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να ενσωματωθούν και στον προϋπολογισμό του 2017 για την τρίτη μεταφορά. Της εξωτερικής δράσης. Ο εισηγητής να απαντήσει. Μπορώ να σας πω για τις δύο πρώτες, ε, ναι, έχετε εκφράσει την άποψή σας για τις δύο πρώτες μεταφορές. Έχει να απαντήσει κάτι ο εισηγητή, όχι. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι επειδή είναι μικρά τα ποσά, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Επιτροπή Προπολογισμών εγκρίνει αυτέ τι δύο μεταφορέ. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα, κύριε εισηγητά, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Πρόκειται κύριε Πρόεδρε για μεταφορά 1.349.000 ευρώ από το τίτλο 2 για τα ενίκια σε τρεις ε, θέσεις 2030 ε, για τα γραφεία γιατί είναι πολύ μεγαλύτεροι λογαριασμοί 2233 διοργανική συνεργασία. Δεν γνωρίζω πολύ καλά το μηχανισμό. Ζητείτε μια αύξηση 1,1 εκατομμυρίου ευρώ ε, για, τις, ε, για την δημιουργία, για την παραγωγή ε, λεσέπασε, όπως επίσης και για τις αποστολές περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Πρόκειται για αμοιβή ε, του προσωπικού της ΕΙΕΔ, δεν κατάλαβα πολύ καλά. Και όσον αφορά το 2.236, επειδή η υπηρεσία ε, νομικών υποθέσεων χρειάζεται περισσότερους νομικούς για την προστασία ενάντια στον κίνδυνο ε, αμαύρωσης της του και ε, της οικονομικής του κατάστασης. Τι να σας πω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. 111 χιλιάδες 111 ευρώ. 111.000 λοιπόν να ζητά κανείς ε, για τέτοιου είδους θέματα μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να το θέσω το ερώτημα και να ακούσω την απάντηση. Κύριε Φρέζα, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κοιτάξτε, απαντώ όσον αφορά το τμήμα που αφορά τα λεσέ ε, που είναι τα νέα ε, λεσέπασε της ε, Επιτροπής για τη διαχείριση φακέλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το κάνει και για λογαριασμό της ΕΕΔ και θα είναι το βασικό γραφείο πληρωμών που θα ασχολείται με την οικονομική κάλυψη των αποστολών της Έτσι υπάρχει κάποιο κέρδος σε αποδοτικότητα. για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν σημαίνει επιπρόσθετη δουλειά λόγω της υπηρεσίας που παρέχεται στο προσωπικό της ΕΕΔ και ε, υπάρχει μια διοικητική, διοικητικού επίπεδου συμφωνία μεταξύ των δύο οργάνων όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει το λογαριασμό στις υπηρεσίες ΕΙΕΔ ε, ώστε να είναι κάπως πιο αποτελεσματική η διαχείριση σε σχέση με τώρα. Μάλιστα, κύριε Σιγητά. Ένα ερώτημα να θέσω και πάλι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε απλώς το τις τιμές ε, των υπηρεσιών που παρέχει για τα νέα αυτά λεσέ πασέ όπως επίσης ε, και για το σύστημα αποστολών εσείς αυξήσατε δηλαδή τις τιμές σας ή άλλαξε κάτι άλλο Ο κύριος Φρέζα Κοιτάξτε, όταν ετοιμάσαμε τον προϋπολογισμό του 2016 ε, δεν ε, ίσχυε ακόμη αυτή η συμφωνία που, ανέβασα προηγούμε, που ανέφερα προηγουμένως. Υπήρξε μια αύξηση των πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενέγραψε στον προϋπολογισμό της ε, στο πλαίσιο για, τη λεσέπασε, για τα λεσέπασε για, το προσωπικό του και για τις αποστολές, αλλά δεν ζήτησε τις, πιστώσει πιστώσεις ε, για τα λεσέπασε για τη διαχείριση των αποστολών του προσωπικού της ΕΙΕΔ. Και το έμβασμα τώρα που ε, ζητούμε σκοπό έχει, η υποθέτω, να καλύψει αυτό το κόστος. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που είχε προβλεφθεί για την ΕΕ το 2016. Κύριε Μανκά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άλλο ένα ερώτημα. μετά βάσει των πληροφοριών αυτών έχει προκύψει μια νέα ανάγκη οικονομική για την ε, Μάλλον κάτι τέτοιο, ναι, για εξοπλισμό γραφείου, αλλά αυτό το ποσό είναι πιο ψηλό από ό,τι προβλεπόταν. Υπάρχει κάποια εξήγηση για όλα αυτά τα θέματα. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί γίνεται κάτι τέτοιο. Και για την περίπτωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εγώ θα ήθελα μια απάντηση από την Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λιγότεροι μεταφραστές μέσω του ίντερνετ και τώρα πρέπει να πληρώνουμε περισσότερο για εξωτερικές υπηρεσίες. Θα διατηρηθεί αυτή η κατάσταση ή θα υπάρξουν νέοι υπάλληλοι οι οποίοι θα προσληφθούν για την μετάφραση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μονκά εγώ είμαι ο διευθυντή του προπολογισμού ε, της, ε, του δικαστηρίου, με τη μείωση του προσωπικού, δεν σημαίνει ότι απολύσαμε ε, νομομαθείς ε, γλωσσομαθείς νομικούς. απλώς υπήρξε μια προσπάθεια περικοπών σε όλα τα όργανα και αυτό υποχρέωσε το δικαστήριο να αλλάξει την πολιτική του γιατί η εσωτερική του ικανότητα μετάφρασης με τη μείωση των ε, ε, του προσωπικού του, ε, επειδή βρισκόμαστε σε πλαίσιο μείωσης των δαπανών μας, μας, δίνει την, μας υποχρεώνει να αλλάξουμε την πολιτική μας, γιατί αυξάνεται όγκος της μετάφρασης και πρέπει ένα τμήμα να το κάνουμε εξωτερική ανάθεση, ένα μεγαλύτερο τμήμα. Υπάρχει λοιπόν μια αλλαγή πολιτικής, ε, Είχαμε συνηθίσει, υπήρχε τέλος πάντων ένα ποσοστό εξωτερικής ανάθεσης γύρω στα 25% και τώρα αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί. Επομένως αυξάνουμε και τον προϋπολογισμό των ε, freelance ε, μεταφραστών. Το 2015 πάλι το κάναμε με ένα συμπληρωματικό ποσό 550.000. Φέτος είναι ε, πιο μεγάλο το ποσό γιατί αυξάνεται και ο όγκος της μετάφρασης και θέλουμε να ε, συνάδει αυτό με την αύξηση του προπολογισμού για τους freelance μεταφραστές που θα, θα προτείνουμε για την επόμενη χρονιά. Μειώνουμε, ε, σεβόμαστε την μείωση του 5% που κάνει οικονομία βέβαια ως πολιτική, αλλά σε μερικές περιπτώσεις ε, είμαστε ε, υποχρεωμένοι να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για τις ε, υπηρεσίες, νομίζω. Κοιτάξτε, δεν μου φαίνεται ότι είναι και η καλύτερη δυνατή διαχείριση. Απλώς και μόνο επειδή έχουμε αποφασίσει κάτι επισήμως ε, να ε, κάνουμε συνεχώς εξωτερική ανάθεση μου φαίνεται λίγο περίεργο. Μιλήσατε επίσης και για έναν κίνδυνο αμάβρωσης φήμης. Ναι, Κοιτάξτε, ένα ερώτημα είναι αυτό που θέλω να θέσω, γιατί ζητάμε ενίσχυση για τις ε, αποζημιώσεις, για την προστασία έναντι του κινδύνου αμάβρωσης φήμης του πώς είναι δυνατόν ε, εκ των προτέρων να πούμε ότι θα υπάρξουν τέτοιου είδους ε, ε, προσβολές της φήμης τέλος πάντων. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, υπάρχει κάτι που έχω χάσει, δεν έχω καταλάβει. Μου φαίνεται πραγματικά πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Κύριε Φρεζά, μπορείτε να μας πείτε για τη φήμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάξτε, είναι ένα εμβάσμα που αφορά την ΕΙΕΔ. Είναι ένα αυτόνομο, ναι, κοιτάξτε, αλλά το θέμα, το θέμα είναι πώς δηλαδή θα μαζέψουμε λεφτά στην ΕΙΕΔ και αυτό εσείς το λέτε μεταφορά. Ναι, θα σας εξηγήσω για τα άρθρα που έχω να κάνουν με το καθεστώς. Όχι, αυτό είναι άλλο, λέει ο κύριο Δεπρέ. Όχι, όχι. Τα άρθρα που έχουν να κάνουν με το καθεστώς ε, είναι η νομική ενίσχυση όσον αφορά τις καταγγελίε ε, του προσωπικού. Άρθρο 2233. Εγώ μιλάω τώρα για το 2236 τώρα. Για το 2236 θέλω να μου πείτε. Μήπως θέλετε να το συζητήσουμε την, στην επόμενη συνεδρίαση. Κοιτάξτε, δεν λέω ότι είναι και τρομερά σοβαρό ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτή η προστασία έναντι, στη, έναντι της προσβολής της φήμης της ε, Επιτροπής. Δεν είναι δεσπό, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Ο κύριο Φρέζα, λοιπόν, αν, δεν αν συμφωνείτε, εγώ δεσμεύομαι να σα στείλω τις περαιτέρω πληροφορίε γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή την απάντηση, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή στο ερώτημα. Ε, μπορώ να σας ε, υποβάλω την απάντησή μου, βέβαια, γραπτό. Εκτός μικροφώνου, τα σχόλια. Πρόεδρος, κοιτάξτε, για τα δύο πρώτα μπορούμε να αποφασίσουμε. 2.230 ε, και 2.230 ε, και 2.233 και το 2.236 να το αναβάλουμε για την επόμενη φορά. Δεν χρειάζεται για τα δύο πρώτα να ψηφίσουμε δεδομένων των ποσών για τα οποία πρόκειται. Αν, ε, αν δεν διαφωνείτε, προτείνω αυτά τα δύο πρώτα... Με, α, μαζί μαζί πρέπει να τα ψηφίσουμε όλα. Ε, τότε όλα θα τα αναβάλουμε για την επόμενη ε, φορά. Κυρία Γολμέιερ. της, ε, του θεματολογίου της μετανάστευσης θα υπάρξουν νέες αρμοδιότητες για το ΕΑΣΟ. Αυτό θα σημαίνει ότι θα χρειαστεί και περαιτέρω προσωπικό και χρειάζεται και περαιτέρω συντονισμό του προσωπικού που εργάζεται στα hot spots μετά από το 2012. Το ΕΑΣΟ έχει ήδη ένα κτίριο στο οποίο δράζεται στο, στην, στο λιμένα της ε, Βαλέτα. Είναι μια πολύ ε, θέση η οποία μπορεί να καλή θέση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ΕΑΣΟ γιατί αποφάσισε το Συμβούλιο ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι αυτό το γραφείο στο λιμένα της ε, Βαλέτα. Είναι τρία συγκροτήματα. Το, κτήριο, το συγκρότημα των κτηρίων είναι σε τρία κομμάτια και τα αυτά έχουν το ΕΑΣΟ με 95 ε, μέλη του προσωπικού και κάποια άλλα τμήματα του κτηρίου χρησιμοποιούνται για συνεδρίες. Υπάρχει τώρα και το νέο το κτίριο ΣΕ, το οποίο θα έχει και επιπλέον κτίρια, μεγαλύτερα κτίρια και θα υπάρχει και ένα κέντρο εποπτείας και μία ε, καντίνα όπως και αίθουσες συνεδριάσεων και Υπάρχει ένα πρόσθετο, μια πρόσθετη έκταση 450 τετραγωνικών μέτρων. λοιπόν, το κόστος μαζί με το κόστος της μίσθωσης και τα λοιπά είναι 1,58 εκατομμύρια. Το... Και στην περίπτωση του ΕΑΣΟ είναι υψηλότερο το κόστος της μίσθωσης γιατί υπολογίστε εκεί το σύνολο του κτηρίου σε βάση τετραγωνικών αλλά αυτό περιλαμβάνει και τις προσβάσεις λοιπά. Αλλά φυσικά η Βαλέτα δεν είναι το φθηνότερο μέρος για να υπάρχει ένα ε, κτίριο αυτού του είδους, γιατί όλη μέρα στο έχει εξυγχρονιστεί και είναι ακριβά τα κτίρια αυτά. Υπάρχει και το κτίριο αυτό λοιπόν το οποίο θα, ένα νέο κτίριο το οποίο θα έχει χώρο για 50 μέλη του προσωπικού και επιπλέον θα υπάρχουν οι αίθουσες συνεδριάσουν το κόστος είναι περίπου 180 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σε ορισμένε περιπτώσει ξεπερνάει τα 200 ε, ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Το συνολικό κόστος για τα κτίρια αυτά μαζί με την ε, τα λοιπά είναι περίπου 1,679 εκατομμύρια. Έχουμε πρόσθετο κόστος 2,86 ε, εκατομμυρίων. Έχουμε το πάρκινγκ λοιπόν, έχουμε 34 πρόσθετες ε, θέσεις παρκαρίσματος και το κτίριο αυτό ανήκει στην μαλτεζική κυβέρνηση οι 34 αυτές θέσεις κοστίζουν 610 ευρώ η μία και αυτό το βρίσκω κάπως ε, αξιοσημείωτο. Καταλήγουμε λοιπόν σε ένα συνολικό ποσό 2,9 εκατομμυρίων το χρόνο. Βέβαια, με τον τρόπο αυτό το ΕΑΣΟ έχει ε, οδηγήσει σε συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών. Θα ήταν πιο φτηνά άλλα κτίρια ενδεχομένω, αλλά άμα σκεφτούμε όλες αυτές τις ε, μετακινήσεις που θα χρειαζόταν, τελικά δεν είναι τόσο ακριβό. Δεν ε, μας ζητά η κυβέρνηση της Μάλτας να υπάρξει τη μαθηνική αναπροσαρμογή στο μίστομα και νομίζω ότι τα κτίρια είναι ήδη έτοιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την συνολική αυτή ενέργεια και το μόνο το οποίο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι ότι ίσως είναι υπερβολικό το τίμημα για τις ε, θέσεις παρκαρίσματος, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την ε, πρόταση αυτή και δεν πρέπει να υπερδραματοποιήσουμε την κατάσταση και για την επόμενη φορά θα ήθελα να έχουμε μια καλύτερη πληροφόρηση εκ των προτέρων και να έχουμε τις σωστές πληροφορίες γιατί την τελευταία φορά είχαμε εγκρίνει επί τη βάση λαθασμένων στοιχείων. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό με μια αποκεντρωμένη υπηρεσία και ζητώ από την Κομισιόν να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Η ΕΑΣΟ έχει βέβαια πολλά καθήκοντα που πρέπει να αντιμετωπίσει, αλλά ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε την Κομισιόν να συλλέγει καλύτερα τα στοιχεία, ώστε να μην χρειάζεται η ΕΑΣΟ να ασχολείται με την κριτήριακή της πολιτική, αλλά συγκεντρώνει τις προσπάθειές της στην Ελλάδα και την Ιταλία στα hot spots. Βέβαια, δεν είναι καλό για το ίδιο κτίριο να υπάρχει διαφορά στην ε, εκτίμηση κατά 300.000. Γι' αυτό παρακαλώ την Κομισιόν να δώσει περισσότερη αρρωγή για τα κτηριακά θέματα στους αποκεντρωμένους φορείς. Κατά τα άλλα, νομίζω δεν θέλουμε να θέσουμε την ΕΑΣΟ σε κατάσταση δυσκολίας γιατί δεν θα βρούμε και κάτι πολύ πιο φθηνότερο. Δεν θέλετε λοιπόν να αναβάλουμε τη λήψη απόφασης, περιμένοντας τις συμπληρωματικές ε, πληροφορίες, τις οποίες ζητήσατε αλλά δεν έχετε. Λέτε να ψηφίσουμε τώρα. Συμφωνεί η Κομισιόν, η Επιτροπή μας μάλλον. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Δεν υπάρχει κανένα κατά. Η απόφαση είναι λιμενη και θα ζητήσουμε από την ΕΑΣΟ με τη βοήθεια της Κομισιόν να μας αναφέρει τι ακριβώς γίνεται με το κόστος του πάρκινγκ. Και ίσως μπορούμε να απευθυνθούμε κατευθείαν και στην ε, μαλτέζικη κυβέρνηση αν δεν πάρουμε πληροφορίες από την ΕΑΣΟ. Πράγματι, θα γράψουμε ένα γράμμα διαμαρτυρίας και θα παραλάβουμε το ένμεσο. Δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε, γιατί στα διάφορα ο Γενικός Συγητής του Προϋπολογισμού έχει να θέσει ένα ερώτημα στην Κομισιόν για ένα αυτόνομο, μια αυτόνομη μεταφορά πιστώσεων 18 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για κάτι το οποίο παρακάμπτει την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αυτό είναι νόμιμο, αλλά αν γίνεται με, με, με χρήση διακριτικής ευχέρειας, θα θίξει την διαφάνεια και έτσι η Κομισιόν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να περνά από το παράθυρο αυτό που δεν μπορεί να περάσει από την πόρτα. Πρόκειται για μια μεταφορά πιστώσεων 18 εκατομμυρίων στο μέσο γειτονίας προς το μέσο προενταξιακού χαρακτήρα για να χρηματοδοτηθεί η ενέργεια για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Μπορεί να μας πει βέβαια η Κομισιόν ότι ξέραμε ότι το μέσο γειτονίας θα πρέπει να συμβάλλει και στη χρηματοδότηση των ενεργειών για τους πρόσφυγες. Ποτέ μας δεν μας είπε ποιο θα ήταν το ποσό. Ποτέ, δεν, ποτέ δεν είπε ότι θα γινόταν με μια αυτόνομη μεταφορά πιστώσεων. Νομίζω ότι μια σωστή λύση για το θέμα αυτό είναι να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο. Αυτή η αυτόνομη λοιπόν μεταφορά πιστώσεων είναι εφικτή μόνο χάρη στις τροπολογίες που κάναμε στη διαδικασία συνδιαλέγης. Είναι λοιπόν αποτέλεσμα και της θέσης του Κοινοβουλίου. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει θέμα, αλλά απλώ το αναφέρω και αυτό το οποίο θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιό είναι να μας πληροφορείτε για αυτά τα 18 εκατομμύρια. θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποια ψήγματα πληροφορίας, κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματά σας για τα σχεδόν 8 εκατομμύρια που αφορούν τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Αφρικής και της γειτονίας μας. περιλαμβάνονται εδώ πηγές χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Τα κονδύλια τα οποία περνούν από, το, τα καταπιστεύματα και από τις υποσχέσεις των δωρητών της συνδιάσκεψης του Λονδίνου και επίσης την μακροοικονομική αρρωγή. Όλα αυτά καταλήγουν σε, 8 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο 8 ετών και για τα καταπιστεύματα περιλαμβάνουν το ποσό που περιμένουμε ότι τα κάτι μελη θα συνεισφέρουν ως ισόποσο του ποσού που δίνει ο προϋπολογισμός ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Για τα 8 δισεκατομμύρια λοιπόν Ούτως έχουν τα πράγματα. Για το είδος των ε, ε των ε, χρήσεων που θα δοθούν σε αυτά τα χρήματα, όλα αυτά εξαρτώνται από τις συμφωνίες εταιρικού χαρακτήρα με τις χώρες προτεραιότητες που αναφέρονται στην ανακοίνωσή μας και φυσικά εξαρτώνται και από τη μορφή που θα πάρει το μείγμα μέσων που θα αφορά τις, ε, ε, υποστηρίξεις προς τα, τις ε, επιδοτήσεις μάλλον προς τα δάνεια που θα δοθούν. Για το σχέδιο επενδύσεων για την Αφρική όπως αναφέρθηκε η Κομισιόν θα έρθει στις 6 Σεπτεμβρίου με πιο εξειδικευμένες προτάσεις. Η πριτανεύουσα ιδέα είναι να υπάρξει μια δυνατότητα να συμμετάσχει περισσότερο το Ταμείο αυτό για να υπάρξουν και ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες θα προσθεθούν στην δημόσια υποστήριξη στις χώρες της Αφρικής και τις χώρες της γειτονίας για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε που κάνουν τους πολίτες των χωρών αυτών να μεταναστεύουν προς την Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικός ρόλος ο οποίος μπορεί να διαδραματιστεί για πηγές χρηματοδότησης ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Υπάρχει ρόλος για τα κράτη-μέλη τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν διμερή βοήθεια. Υπάρχει ένας δυνητικός ρόλος επίσης για τις ε, αναπτυξιακές ε, τράπεζες και του αναπτυξιακού αναπτυξιακούς φορείς οι οποίοι δανειοδοτούν τέτοιου είδου ενέργειες ανάπτυξης είτε σε διεθνές επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο και επομένως οι προτάσεις αυτές θα έχουν σαν στόχο να συναθρήσουν και να συναρμόσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Και οι νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα έρθουν εν καιρό, ιδίως για τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας επενδύσεων, θα έρθουν στο μέλλον, αν δεν έχω αφήσει με ένα συγκεκριμένο συγκεκριμένο χρόνο-διάγραμμα για να σας πω περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φρέζα για όλες αυτές τις διευκρινήσεις. Μήπως θα μπορούσατε σε σχέση με το πρώτο ερώτημα των 8 δισεκατομμυρίων να μας στείλετε ένα έγγραφο για να ξέρουμε ακριβώς πώς, ε, ποιες είναι οι διάφορες ε, ε, εισφορές για να φτάσουμε τα 8 δισεκατομμύρια και επίσης πώς ε, ε, χρησιμοποιούνται αυτά τα 8 δισεκατομμύρια, πώς κατανέμονται ετησίως. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις αυτές. Μήπως υπάρχουν άλλα θέματα υπό τα διάφορα. Όχι. Άρα, μπορούμε να κηρύξουμε το πέρας της συνεδρίαση αυτής. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας.